Καλημέρα κύριε και κύριοι. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά την πρωινή μα συνεδρία στην δεύτερη μέρα. Second day. Uh, <clears throat> uh Λοιπόν, Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα, διαπραγματεύσεις για την TTIP, διατλαντική εταιρική σχέση δηλαδή στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. Ε, καλωσορίζω τον τμήματάρχη ε, για ε, αρμόδια αυτά τα θέματα, τον κύριο Λουκ Κέβιν από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Σωστά το είπα το όνομά σας. Καταπληκτικά. Και δεν ρώτησα και κανένα, το βρήκα μόνος μου. Λοιπόν, θα μπορούσατε σύντομα να μας ενημερώσετε για το πώς έχει η κατάσταση των διαπραγματεύσεων και πώς προχωρούν. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας, τα θέματα της ενέργειας και των πρώτων υλών, που είναι και η αρμοδιότητά σας. Και αν υπάρχει κανένα σχέδιο να συμπεριληφθεί ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια. Μετά έχουμε τα ρυθμιστικά θέματα, οι ευκαιρίε ε, επίση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας ενδιαφέρουν. Κατά το 12ο γύρο διαπραγματεύσεων που διεξήχθη στις Βρυξέλλε από τις 22 μέχρι τι 26 ε, Φεβρουαρίου εστότο έτους. Σίγουρα ε, θα αναφέρετε πολλά από τα θέματα αυτά. Θα τα συζητήσετε και έχει σημασία να γνωρίζουμε εμεί τι τρέχει εκεί. Αυτά. Θα θέλαμε και ένα γενικότερο σχόλιο για το πώς βλέπει το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων και τις προγραμματισμένες επόμενες διαπραγματεύσεις και τους σχετικούς γύρους. Έτσι πώς θα συνεχιστεί από εδώ και μπρος η διαπραγμάτευση, κυρίως, διότι ε, τα τέλη του έτους ξέρουμε ότι έχουν προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και είναι λίγο πιο δύσκολη φετινή χρονιά ως εκλογική. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Θα ξεκινήσω με μια γενική επισκόπηση του γύρου του περασμένου μηνός και θα εστιαστώ λίγο περισσότερο σε θέματα ενεργειακά και πρώτων Όσον αφορά την γενική κατάσταση και προοπτικές, πήγαμε καλά τον προηγούμενο μήνα, εστιαστήκαμε επί, δύο, επί τριών πυλώνων, ρυθμιστικό και τον πυλώνα των κανόνων. Όπως ξέρετε ήταν επικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ της ε, ε, Επιτρόπου Βάλστρομ και των Αμερικανών ομολόγων. Τώρα το ρυθμιστικό πλαίσιο, προχωρήσαμε καλά για ρυθμιστικές πρακτικές και ρυθμιστική συνεργασία και επί των δύο κεφαλαίων λάβαμε πρώτη πρόταση τον ΗΠΑ για την συνεργασία για τα ρυθμιστικά θέματα. Θέλουμε να εκτιμάσουμε ένα κείμενο για τις προτάσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ενώσης μέχρι τέλος ε, Ιουλίου θα είναι έτοιμο το κείμενο. Τεχνική φραγμή στο εμπόριο. Η προσέγγιση έγινε πιο συμβατή πλησιάσαμε σε κάποιους τομείς και ιδιαίτερους κανόνες όπως για τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα αυτοκίνητα, για τα SPS, για τα φυτογενομικά, τους κανόνες. Εκεί η πρόοδος ήταν μικρότερη. Για, ως, για τους κανόνες τα πράγματα ήταν πιο ανάμεικτα από ότι για το ρυθμιστικό προχωρήσαμε την έρευνα και ανταγωνισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα κλείσει το κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες σύντομα. Ε, ελπίζουμε κάποια κρεμή ζητήματα απομένουν μόνο. Πολύ λίγα. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλάξαμε ταχύτητα. Η ΕΠΑ έκανε προτάσεις όσον αφορά τα εργασιακά και το περιβάλλον. Η πρότασή τους νομίζω ότι εμπνέεται κατά πολύ από την άλλη συμφωνία ε, του Ειρηνικού εμπνέεται πολύ από αυτή, αλλά είναι καλό που υπάρχουν αυτές οι επαφές επί το επικειμένου με τη ΣΥΠΑ όσον αφορά στους άλλους κανόνες που μας ενδιαφέρουν, ενέργεια και πρώτες ύλες και επιδοτήσεις, κρατικές ενισχύσεις της επιχειρήσεις, εκεί προχωρήσαμε λιγότερο και για πρώτη φορά κουβεντιάσαμε για την προστασία των επενδύσεων. Η συμφωνία του Καναδά, το ΣΥΤΑ, είναι σημαντική ε, σημαντικό επίτευγμα, θα έχει επιπτώσεις στη Ουάσιγκτον. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές όμως μεταξύ των θέσεών μας και πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις της επενδύσεις θα ολοκληρωθούν μόνο στο τέλος των διαπραγματεύσεων γιατί είναι δύσκολο κεφάλαιο, πολύ δύσκολο. Τέλος, εξίσου σημαντικό πρόβαση στην αγορά, λίγη πρόοδος επετεύθη, αλλά σε αυτό το γύρο δεν ήταν και στο επίκεντρο της προσοχής μας. Για τις κρατικές προμήθειες λάβαμε πρώτη πρόταση των ΙΠΑ, μετά το γύρο τρέχουμε με την προσφορά και δεν πιστεύουμε ότι θα επιτρέψει να ολοκληρώσουμε το θέμα για τις κρατικές προμήθειες. Είναι σημαντικό επιθετικό συμφέρον τον είπα αυτό, ε, το, της Ευρωπαϊκής Ενώσης, συγγνώμη. Όσον αφορά τις υπηρεσίες είναι δυσχερείς οι συζητήσεις. Στόχος είναι οι κρατικές προμήθειες και υπηρεσίες ε, να οριμάσουν ως θέμα, όπως και για τους δασμούς, στο επίπεδο των δασμών. Για το επόμενο βήμα τώρα, θέλουμε και μπορούμε να ολοκληρώσουμε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Ομπάμα αν πετύχουμε σε όλους τους τομείς των διαπραγματεύσεων συγκρίσιμη πρόοδο. Απομένει να δούμε σε ποιο βαθμό οι ΙΠΑ μπορούν να συνομιλήσουν μαζί μας ενώ ταυτόχρονα έχουν και το θέμα της κυρώσης της συμφωνίας του ελληνικού. Ανεξάρτητα από την ιστορική πολιτική των ΙΠΑ, πολλή τεχνική δουλειά θα πρέπει να γίνει. Έχουμε τον επόμενο γύρο που θα γίνει στη ΣΥΠΑ 25 με 29 Απριλίου αυτή την εβδομάδα και θα γίνει και άλλος γύρος που έχει προγραμματιστεί ήδη και θα λάβει χώρα τον Ιούλιο εν τω μεταξύ θα γίνει πολλή δουλειά άρα θέλουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται όσον αφορά τα κείμενα και μέχρι το καλοκαίρι να καταλήξουμε σε κάποια κείμενα το, το σωστό TTP να είναι έτοιμο για συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο βέβαια τα θέματα Η ΕΠΑ δεν θα μειώσουν φιλοδοξίες για τη Γεωργία αλλά αυτό θα πρέπει επίσης να βρει κάποιο αντάλλαγμα και η εξολόγησή μας παραμένει μια φιλόδοξη συμφωνία που θα είναι ευκολότερο να περάσει από ότι ένα TTP light, αν επιτρέπεται αυτή την έκφραση. Τώρα προχωρώντας στο θέμα της ενεργείας και των πρώτων υλών και το σχετικό κεφάλαιο αυτό που ζητήσατε, στο τελευταίο γύρο Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε επικειμένου, οι Αμερικανοί δεν ήταν έτοιμοι να υποβάλουν προτάσεις κειμένου και λυπούμεθα γι' αυτό. Ανταλλάξαν πληροφορίες όμως το γύρο αυτό περί θεμάτων όπως πρώτες ύλες και ενέργεια και κυρίως για την ενέργεια. Παρουσιάσαμε την όλη κατάσταση της Ενεργειακής Ενώσεως και οι δύο πλευρές συνέκριναν τα αποτελέσματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων με το Βιετνάμ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη συμφωνία του ειρηνικού πλευράς ΙΠΑ. Επίσης ακούσαμε εξηγήσει από τις ΙΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή της ανάκλησης της απαγόρευσης εξαγωγής πετρελαίου που ενέκρινε πριν από μερικές εβδομάδες το Κογκρέσο. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι είμαστε έτοιμοι για επικοδομητικές συζητήσεις για τις σχέσεις μεταξύ ενδεχομένων διατάξεων για τις πρώτες ύλες που συζητούνται και σε άλλα κεφάλαια όπως το εμπόριο αγαθών, εξαγωγική τιμολόγηση, εξαγωγική περιορισμή. Είναι ένα θέμα αυτό διαφωνίας με τη ΣΥΠΑ. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται ειδικό ενεργειακό κεφάλαιο, διότι πιστεύουν ότι αυτά που ζητούμε στο ενεργειακό κεφάλαιο καλύπτονται από οριζόντιες διατάξεις. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Πιστεύουμε ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία να έχουμε ένα ξεχωριστό ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια Λοιπόν, ολοκληρώνουμε λοιπόν πρόταση κειμένου, η οποία θα υποβληθεί σύντομα, ίσως να μην υποβληθεί έγκαιρα για να διεξαχθούν συζητήσει με βάση το κείμενο για ενέργεια και πρώτες ύλες στον επόμενο γύρο, τον Απρίλιο, λόγω εσωτερικών διαβουλεύσεων που απαιτούνται, αλλά σίγουρα το αργότερο στο γύρο του Ιουλίου το κείμενο θα είναι έτοιμο και πολύ σύντομα θα υποβάλουμε πρόταση με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου βέβαια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις επί του θέματος. Θα παρακαλούσα την κυρία Ντάρλινγκ να πάρει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και Ντελίν για την ε, ενημέρωση. Όπως σας έλεγα, ε, είμαι ένα πληρωματικό μέλος εδώ στην Ίντα, είμαι πλήρες μέλος. Άκουσα την πλήρη παρουσίαση στις αρχές της εβδομάδας από τον αναπληρωτή επικεφαλής της διαπραγμάτευσης. Και σε αυτή τη συνάντηση μας παρουσίασε όλη την πρόοδο. Έχω τρεις ερωτήσεις. Αφορούν ενέργεια, πρώτες ύλες και βιομηχανία, σχετικούς ε, τομείς στην συνάντηση αυτή την εβδομάδα μας είπε ότι είμαστε εν το μέσο του ενδιαμέσου παιχνιδιού αν θέλετε και είναι τακτική του διαπραγματευτή να λέει κάτι χωρίς να εξηγεί ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Τουλάχιστον το καταλάβουν οι απλοί άνθρωποι εκεί που ότι στόχος θα ήταν να εξασφαλίσουμε ένα κείμενο μέχρι το καλοκαίρι και το δεύτερο εξάμεινο του 2016 να επεξεργαστούμε το τελικό στάδιο του TTIP. Λοιπόν, αυτό το χρονοδιάγραμμα, έχοντας αυτό υπόψη, Πού είναι τα κεφάλαια για ενέργεια, τηλεπικοινωνία, ψηφιακή ενιαία αγορά, παράλληλα με την αυτοκινητοβιομηχανία. Πού είναι στο μέσο της ε, διαδρομής. Είναι στοιχεία που θα πάνε στην τελική φάση. Μας δίνετε μια εικόνα. Αναφερθήκατε επίσης σε αυτόν τον όρο που ακούμε του T.T. Lite που συνεχώς αναφέρεται περισσότερο και πιθανότατα να έχουμε μια πιο πρώιμη συμφωνία όπου είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσουν επί λιγότερο πλήρους αλλά και λιγότερο επιμάχου συμφωνίας που θα εστιάζονται στην ρυθμιστική σύγκληση περισσότερο και υπάρχει κάποια άποψη ότι η επίσκεψη του Ομπάμα τον Απρίλιο ίσως θα επηρεάσει την κατάσταση και να επιτευχθεί συμφωνία τότε στην Ευρώπη. Τώρα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν τέτοια συμφωνία τελικά συναυθεί, τι σημαίνει αυτό για την ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και την αυτοκινητοβιομηχανία, του σχετικού τομεί. Αυτά τα κεφάλαια θα συμπεριληφθούν σε αυτή την αρχική συμφωνία, σε μια πρώιμη συμφωνία. Και ποιε θα είναι οι συνέπειε αν συμπεριληφθούν αυτοί οι τομεί. Τρίτη ερώτηση. Ε, μία που προσπαθούσα να την προωθήσω στο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστια προγράμματα ερευνητικά με πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και αυτή είναι στην πρώτη γραμμή για την καινοτομία, για να μέσα ενεργειακή απόδοση και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών και πρασίνων τεχνολογιών. Στις συζητήσεις για την ενέργεια και τις πρώτες ύλε, υπάρχει κάποια συζήτηση, δηλαδή πώς μπορούμε και εμεί να καταβάλουμε κοινέ προσπάθειε από αυτού, κυρίως μετά την COP των Παρισίων πέρσι, ούτω ώστε να καταβάλουμε κοινέ προσπάθειες που πλευρά ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά την ενεργειακή τεχνολογία, την ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες, κάτι που θα έχει έναν ε, αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δερμό, Πράσινος, παρακαλώ. Okay. Στο Παρίσι ε, έγινε η διάσκεψη κορυφής για το κλίμα. Πώς άλλαξε τη θέση της Ευρώπης για την ενέργεια. Ιδιαίτερα για την υδρορογμάτωση και το σχιστολιθικό αέριο. Ή δεν το συζητάτε καν αυτό. Είναι αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Θα τα ξαναπώ. How did, uh, αγγλικά τώρα. Πώς επηρέασε το ε, αποτέλεσμα της διάσκεψης ε, των Παρισίων για το κλίμα και πώς άλλαξε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως δεν έχουμε αλλάξει θέση για αυτό το θέμα. Ε, Η κυρία Λόπες από την ΚΟΕ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που γίνεται καταρχήν αυτή η συζήτηση. Φοβάμαι πως το λίγο που κερδίσαμε εδώ στη διαφάνεια το χάσαμε ε, με την επαλή, σε επίπεδο επαλήθευσης περιεχομένου, για παράδειγμα. Η Κομισιόν κάνει μια προσπάθεια την πρότασή της να την υποβάλει πριν τις διαπραγματεύσεις, σαν να πρόκειται για μεγάλη βελτίωση χωρίς να κάνει ε, αυτό που έκαναν πολύ γνωστοί νομικοί ε, της Ευρώπης, πως αυτά τα δικαστήρια τα οποία συστήνει ε, αντίκειται στην νομοθεσία που έχουμε στην Ευρώπη και λένε πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν κινδυνεύει. Όμως κινδυνεύει. Και θα σας αναφέρω ότι έγινε με τη Volkswagen μετά από τις επανειλημμένες παραβιάσεις των προτύπων και των κανόνων εκτός επομπών, ε, με συγχωρείτε, παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή μία, ε, μία πρόταση η οποία ε, εκ των υστέρων δικαιολογεί αυτές τις παραβιάσεις. Μα τι είναι αυτή η πρόταση, μία θεσμοθέτηση αυτών των πρακτικών. Δεν θεωρείτε πως εκλείπει η δημοκρατία όταν αφήνουμε στους τεχνικούς τα θέματα αυτά και στις πολυεθνικές να προτείνουν, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τον, τους κανονισμούς που εγκρίνει εδώ το Κοινοβούλιο. Στη χώρα μου ανακοινώθηκε πρόσφατα πως θα κλείσει προσωρινά, θα κλείσει προσωρινά δύο χαλιβουργίες. Δύο. Οι συνάδελφοι και σύντροφοι στη Γαλλία και στην Αγγλία μπορούν ε, να μας δώσουν πολλά παραδείγματα το πόσα καταστρεπτική είναι, καταστρεπτικός είναι ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό για το χάλιβα. Η Κομισιόν πέρσι ε, σε μια μελέτη κατάφερε να αποδείξει πως η ίδια η συμφωνία θα έφερνε μια πτώση στην παραγωγή μετάλλων. Να το ξαναδούμε γιατί έχω την εντύπωση πως η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει πως η πρόσβαση στην αγορά υποδομών στην, στη ΣΥΠΑ θα καλύψει τις ζημιές από ό,τι τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε στο δικό μας βιομηχανία, βιομηχανικό κλάδο. Μα αυτό απλώς θα αυξήσει την ανεργία. Δεν υπάρχει ε, κοινωνική πρόοδος χωρίς βιομηχανία και η συμφωνία δεν αφήνει χώρο για βιομηχανία στην Ευρώπη. Κύριε ναι, πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Ξέρετε, καθυστέρησα γιατί είχε ποτηλιάρισμα εκείνη στο δρόμο για το TTIP. Δεν ήθελα να επανέλθω σε μια βασική έννοια που είναι η έννοια της κυριαρχίας. Μήπως θέλει που σε άλλη ζωή ήμουν φιλόσοφος ή θεολόγος και αισθάνομαι υποχρεωμένος να το κάνω. Ε, κυριαρχία είναι ο ίδιος ο λαός. Και ακόμη και αν ε, πίστευαν κάποιοι ότι υπήρχε κυριαρχία, λέω Θεό, όπως ο Θωμάς ο Ακινάτης, περνούσε μέσω του λαού. Δηλαδή ο λαός την επαλήθευε. Και τώρα θέλουμε, λέει, να κάνουμε μια συνθήκη, την οποία, λέει, δεν τη θέλουν. Μα, ε, και αν ψηφίσατε τώρα, αν αφήνατε τον κόσμο να ψηφίσει, θα το διαπιστώνατε. Και αναρωτιόμαστε και για τις Ηνωμένε Πολιτείε, αν το θέλουν. Ακούμε τι λέει ο Τραμπ και ο Σάντερ. Ποια είναι λοιπόν η δική σα νομιμοποίηση, ε, έτσι ώστε σήμερα να μας δεσμεύσετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη συνθήκη αυτή. Το έχετε αναρωτηθεί αυτό. Γιατί υπάρχει και ένα φυσικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, που προβλέπει και το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Διότι περί αυτού πρόκειται αυτό που κάνετε τώρα. Είναι σχάτη προδοσία. Διαπραγματεύεστε κάτι ενάντια στη βούληση του λαού και ε, αναγκαστικά. Αυτό το θεωρείτε φυσιολογικό και νομίζετε ότι θα σας αφήσει η ιστορία να κάνετε τέτοια πράγματα. Ακόμα και αν περάσει το δικό σας και η συνθήκη αυτή, αυτό θα γίνει. Αυτή είναι η σταγόνα που κάνει το ποτήρι να ξεχυλήσει. Δεν θα επανέλθω στην ουσία, δεν θα επανέλθω στην ουσία. Που μόνο να χάσει έχει η Ευρώπη. Και τα πάντα μάλιστα. Και το γνωρίζετε. Και μας κάνετε να πιστεύουμε το αντίθετο. Γιατί δεν είστε πραγματικά Ευρωπαίοι που θέλετε να εργάζετε υπέρ των λαών της Ευρώπης. Σα ευχαριστώ. Uh, um, uh, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλουάγα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι θέλετε να συζητήσουμε γιατί ε, δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό που διαβάζουμε και η μόνη ενημέρωση που έχουν οι πολίτες σήμερα για θέματα ενεργειακά είναι αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ρωτήσω ε, πώς σχολιάζετε εσείς αυτή την κατάσταση. Επίσης, εμείς θεωρούμε πως η συμφωνία αυτή για τα ενεργειακά ζητήματα έχει ως στόχο ο ανεφοδιασμός σε ορυκτά καύσιμα να ανοίξει και σε εισαγωγές από τη Δύση ε, μέσω της συμφωνίας TTIP έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε τα γεωστρατηγικά μας συμφέροντα και να εξασφαλίζουμε ε, την ασφάλεια του ανεφοδιασμού γιατί από ό,τι κατάλαβα, οι ΙΠΑ στο θέμα αυτό δεν θέλουν να διαπραγματευτούν και νομίζω ότι ε, δεν πρόκειται να εξυπηρετήσουν αυτά τα αιτήματά μας. Άρα λοιπόν, για, μη, ε, για πρόσκοτη με συγχωρείτε πρόσβαση στα, πετρελαϊκές, ε, στα πετρελαϊκά αποθέματα ε, τον είπα τι θα πρέπει εμείς να δώσουμε σε αντάλλαγμα είναι η κοινωνική, τα κοινωνικά δικαιώματα είναι οτιδήποτε άλλο επίσης για το σχιστολιθικό και την ε, επίδραση που θα έχει στο χάρτη της ενέργειας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μου πείτε ε, τι βλέπετε σε αυτή τη συμφωνία για τη ΣΑΕΠ που να ευνοεί τη ΣΑΕΠ στα πλαίσια των στόχων για το 2020. Τι γίνεται με τα αέρια του θερμοκηπίου. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Σκοφόρ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση. Εδώ κάθομαι. Μία σύντομη ερώτηση, γιατί νομίζω το έχουν ήδη θέσει συνάδελφοι. Στο κεφάλαιο που έχουμε ε, για την ενέργεια και για τις πρώτες ύλες, θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν στο κεφάλαιο αυτό. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι καλή συνεργασία για τις ε, ΑΠΕ να δούμε πώς μπορούμε να προκρίνουμε και την ε, έρευνα σε αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ξέρετε ότι εκεί με τη ΣΥΠΑ έχουμε κάποιους περιορισμούς μέσω της νομοθεσίας, προστατεύουν την αγορά τους, έχουν το θέμα με τα αιωλικά πάρκα, οπότε θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς σημαίνει για σας ε, και πώς έχουν ε, λάβει αυτό αυτά τα αιτήματα οι Αμερικανοί, κυρίως για τα πράσινα αιωλικά, ε, για τα πράσινα ενεργειακά πάρκα. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα. Έχουμε 10 εκατομμύρια μικρομεσαίες, δεκάδες εκατομμύρια μικρομεσαίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είδους ε, εξαρτή ενημέρωση θα προτείνετε από τη στιγμή που η συμφωνία ε, μπορεί τελικά να υπογραφεί. Και γιατί θα είναι θετική για την ανταγωνιστικότητα, πώς θα επηρεάσει το οικονομικό μας μέλλον. Επίσης, έχουμε το νέο κεφάλαιο στην ενέργεια. Από τι αποτελείται και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε να ανοίξει ε, για το LNG για παράδειγμα η αγορά των ε, Αμερικάνων. γιατί υπάρχει εδώ και 43 χρόνια, υπήρχε μάλλον μια απαγόρευση για τις εξαγωγές αργού, αλλά ε, θα ήθελα να μου πείτε αν παρόλο που αυτή η νομοθεσία έχει καταργηθεί, εάν ε, για το LNG έχει αλλάξει κάτι ή αν θα το εντάξει εσεί στο κεφάλαιο αυτό, έτσι ώστε να είναι οι ίδιοι οι κανόνες παιχνιδιού για όλους ε, στη σχέση μας με τη ΣΥΠΑ. Διαφορετικά, Η μείωση που έχουμε προτείνει εμείς για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, δεν ξέρω πώς θα συνδυαστεί με τις υποσχέσεις που δώσαν οι Αμερικανοί στο Παρίσι. Και νομίζω δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε με τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ και εσάς κύριε Πρόεδρε και τα αξιότιμα μέλη για τις δηλώσεις ή ερωτήσεις που κάνατε. Να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζετε, εμείς τα θέματα αυτά τα αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα, γιατί προσφέρουν πολλές θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Και πάντα έχουμε κατά νου να έχουμε συγκεκριμένα κεφάλαια που να απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες. Στη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, εμείς αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε ένα σημείο ένα σύστημα με, σημείο, με σημεία επαφής, με μια διαδικτυακή σελίδα ε, που θα αναρτώνται όλοι οι κανονισμοί και οι διατάξεις και αυτά θα δημιουργηθούν ε, και θα πληρωθούν και από τη ΣΥΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το Παρίσι και για την πράσινη ενέργεια. Το έχουμε πολύ στο μυαλό μας και θα συμπεριλάβουμε στο κεφάλαιο το οποίο θα υποβάλουμε ε, πολλούς κανόνες ε, για τη ΑΠΕ, για την ενεργειακή αποδοτικότητα, εκεί θα συμπεριλάβουμε και τη συνεργασία. Ακούσαμε και κάποιες ε, ερωτήσεις ε, για την τεχνική της ρογμάτωσης και εάν θέλει κάποια εταιρεία να προχωρήσει σε τέτοιου είδους τεχνική ε, επεξεργασία, αυτό δεν θα επιτρέπεται μέσα από τις διατάξεις συμφωνίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να έρθουμε σε αντίφαση και σε αντίθεση με τους, με τους κανόνες που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν ε, οι συνάδελφοι εδώ, οι δικοί μου θέλουν κάτι να ε, συμπληρώσουν. Για το LNG έχετε δίκιο. Η απαγόρευση για το αργό έχει αρθεί, αλλά για το LNG όντως υπάρχει ένα σύστημα εξαγωγικών αδειών που είναι αρκετά περίπλοκο και αρκετοί από τους δικούς μας ε, εμπορικούς φορείς δεν έχουν εύκολη πρόσβαση ή καθόλου πρόσβαση σε αυτή την εμπορική σε αυτό, το μερίδιο της αγοράς. Θέλουμε λοιπόν να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και συμφωνούμε απόλυτα πως θα πρέπει σίγουρα η να υπάρχουν διατάξεις που θα έρουν τέτοιου είδους εμπόδια ε, οποίε πολλέ φορέ δεν κάνουν άλλο από τον επιβραδύνουν το εμπόριο. Και νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί και τα συμφέροντα των ΗΠΑ, γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο εμεί επιθυμούμε είναι η, να παρεμβαίνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ ε, με τέτοιου είδου ε, κανόνες. Για την πρώτη ερώτηση, ε, αν θα πω κάτι διαφορετικό από ό,τι είπαν οι συνάδελφοι στην Ίντα, δεν νομίζω. Αν είχα να πω κάτι διαφορετικό, θα με κατηγορούσατε ότι προσπαθούμε να παραπλανήσουμε το κοινοβούλιο. Τώρα για το αν είναι το μεσαίο παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κάποιος που βρίσκεται. Όταν θα αντιδράσουν ε, οι είπα ε, προτάσεις που έχουμε κάνει γραπτά για τα ενεργειακά, θα γνωρίζουμε πόσο δυνηρό είναι για τις ΗΠΑ να τα δεχτούν. Και αυτό θα ορίσει και το χρονοδιάγραμμα για να δούμε πώς μπορούμε να σημειώσουμε. Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τις είπα. Οπότε και για τη συνεργία και, και για τη συνεργασία και ε, για τα ενεργειακά να σας πω πως όντως καταρχήν θα έχουμε για τα προγράμματα συνεργασίας κάποιους συγκεκριμένους κανόνες αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει ε, να, ότι εκεί δεν χρειάζεται να προσφέρουμε κάποια ανταλλάγματα ή παραχωρήσεις. Νομίζω ότι όταν προχωρήσεις στην άρση κάποιων εμποδιών προς το εμπόριο, το κάνεις γιατί και οι δύο πλευρές το επιθυμούν, δεν πιέζουμε κανέναν. το θέμα με την έκθεση για την παραγωγή ε, τη βιομηχανική παραγωγή μετάλλων. Θα ήθελα να τη δω, κυρία Λόπες, δεν την έχω δει. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο και στο συνάδελφο να μιλήσει για την πράσινη ενέργεια. Um, Καλημέρα. Όσον αφορά το κεφάλαιο που θέλουμε να παρουσιάσουμε, δεν συμφωνούμε ακόμα με τη ΣΥΠΑ κατά πόσο θα υπάρξει κεφάλαιο εκρεμεί αυτό. Αν υπάρξει συμφωνία, αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να καλύπτει τα πάντα. Όχι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο να καλύπτει, αλλά και ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και ενεργειακή απόδοση. Και σε αυτό το βαθμό θα προτείνουμε κανόνες που θα προσπαθούν να προωθήσουν τις επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση Καλύτερη συνεργασία για πρότυπα και προδιαγραφές θα θέλουμε να καταφέρουμε. Θέλουμε να προτείνουμε κανόνες για πρόσβαση στο δίκτυο για νεώσουμε πηγές ενέργειας. αυτό ήταν το άλλο ερώτημα που ετέθη. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να περιορίσουμε το περιεχόμενο περαιτέρω που αποτελεί εμπόδιο στο θέμα της ενέργειας και αν θα έχουμε αγαθά και υπηρεσίες πώς θα, τι θα προβλέπετε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ε, για την ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε εκεί και τη συνεργασία στα θέματα της έρευνας, να υπάρχει αυτή η συνιστόσα. Όχι μόνο σε αυτό το τομέα, αλλά και σε αυτό το τομέα να συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. It's, uh, uh the, the next... Uh, Κοιτάξτε, ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί τέλος Απριλίου. Και θα καλέσουμε τον Μάιο ή τον Ιούνιο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενημερωθούμε. Μπορείτε να πείτε πότε προβλέπετε να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Πώς το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτίμηση, λίγο πολύ. Να έχουμε έτσι μια εικόνα για το χρονοδιάγραμμα, όχι σε τάξη ημερών ή μηνών, αλλά έστω ετών. Σε τέτοια κλίμακα μπορείτε να πείτε κάτι. Απάντηση. Δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα. Όλοι γνωρίζουν ότι αν δεν πετύχουμε κάτι φέτος, επειδή οι Αμερικανοί αργούν μέχρι να λειτουργήσει και η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι μέχρι τέλος του έτους, δεν ξέρω, ίσως αρχέ του επομένου έτους, έχω αμφιβολίες. Μαντεύω τώρα. Και δεν θέλω να μαντεύω. Και αν ήμουν καλός στο να μαντεύω θα έκανα άλλη δουλειά. Οι ΙΠΑ έχουν συνάψει συμφωνία με κάποιες χώρες της Ανατολικής Ασίας από ό,τι γνωρίζουμε. Εμείς δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί όπως οι άλλοι. Όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο με τη ΣΥΠΑ, ας περιμένουμε. Εμείς διαπραγματευόμεθα καλύτερα. Λοιπόν, καλή απάντηση αυτή. Το τέλος των συζητήσεων. Ευχαριστώ που μας δώσατε πληροφορίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ως γνωρίζετε, σε ένα 20 λεπτό θα διεξαχθεί η ψηφοφορία και θα σας παρακαλούσα να μείνετε ένα 20 λεπτά ή να πάτε μια βολτίτσα για 20 λεπτά και να τα πούμε εδώ ξανά στις 10 για να ψηφίσουμε. Ε, good morning, good morning, ladies and gentlemen. Good. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. We are as precise at, at the... Λοιπόν, στις 10 η ώρα λοιπόν είχαμε μπλέξει με τον... είχαμε μπλέξει από συνάδελφοι στο σταθμό του Μιντή. Πρώτο σημείο ψηφοφορία. Εκλογή τρίτου αντιπροέδρου της Επιτροπής Ήτρε. Και Έχουμε απαρτία, χρειαζόμαστε 17 ευρωβουλευτές και όλες οι ομάδες ενημέρωσαν ποιοι αντικαθιστούν τα πλήρη μέλη, τα τακτικά μέλη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχάς στο συντονιστή της ΓΚΟΕ, τον κύριο Σιλικιώτη ο οποίος θα παρουσιάσει τον κύριο Κόχλιτσεκ, τον υποψήφιο, τον κύριο Γιάρομιλ Κόχλιτσεκ, για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Συνάδελφε, μισό λεπτό, μισό λεπτό, όλα θα ξεκαθαριστούν. Κύριε Σιλικιώτη. Ε, Mr. Kolicek, Ε, είναι ο ευρωβουλευτής που αντικατάστασε τον συνάδελφο μας ε, Γιάροσλαφ ε, και είναι από τη Τσεχία. Ε, γι' αυτόν τον προτείνομαι για τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου. Ο, ο, ο κύριο Κόλιτσεκ δεν, δεν μπορούσε να ήταν σήμερα παρόν εδώ λόγω άλλων υποχρεώσεων που είχε γιατί αυτή η αντικατάσταση έγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ε, έχουμε στείλει ήδη από πριν επιστολές ε, στον Πρόεδρο ε, και εξηγούσαμε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό προτείνομαι για την Πρόεδρο τον κύριο Κόλιτσεκ. Σα ευχαριστώ πολύ. Έχω λάβει δύο επιστολές. Δύο επιστολές. Τη μία από τη Γενική Γραμματεία της ΓΚΟΕ Λέγοντα ότι ο κύριος Κόχλιτσεκ είναι υποψήφιο όπως είπε και ο κύριος Ηλικιώτης ε, από πλευρά της Νοτικής Αριστεράς και έχω λάβει και μία επιβεβαίωση ότι ο κύριος Κόχλιτσεκ συμφωνεί ε, με την υποψηφιότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έχω λάβει και άλλη επιστολή πιο μακροσκελή ε, του ιδίου, του κύριου Γιάρομιλ Κόχλιτσεκ, που απευθύνεται σε μένα προσωπικά ως πρόεδρος και είπε ότι κολλείεται σήμερα να βρίσκεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Και δεν σημαίνει ότι υποτιμά τη σημασία της εκλογής ή της συνεδρίασης, αλλά από την αρχή του έτους είχε αναλάβει άλλη υποχρέωση και δεν είχε ε, ε, σκεφτεί το ενδεχόμενο ότι από το Φεβρουάριο θα ήταν υποχρεωμένος να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έχει αναλάβει μια πάρα πολύ σοβαρή υποχρέωση, ε, οπότε σήμερα κολλιόταν να παρευρεθεί στην ε, συνεδρίαση. Χθε παρευρισκόταν και προσθέτει ότι επειδή... Είμαι παλαιομοδίτης κάπως και αναλαμβάνω να ε, φέρω σε πέρα στα καθήκοντά μου. Αύριο κολλείομαι και δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. Λέει ορισμένα πράγματα για τις δραστηριότητες του. Πάνω από 23 χρόνια ε, εργαζόταν σε ιαλουργία, χαλιβουργία και σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε ε, πορσελάνη πολυτελείας και είναι επιλογή του η συμμετοχή του στη δική μας επιτροπή. Αυτή είναι λοιπόν η εξήγηση που μας έστειλε ο κύριος ο ίδιος και σας ερωτώ αν έχουμε άλλους υποψηφίους. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για την εκλογή. Δεν βλέπω άλλη υποψηφιότητα, οπότε απουσία άλλης υποψηφιότητος ε, ψηφίζουμε διαβοής. Thank you very Σα ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και προχωρούμε. Συγχαρητήρια παρακαλώ να διαβιβάσετε στον κύριο Κόχλιτσεκ. Εχθέ ήταν όλη μέρα εδώ, σήμερα έχει άλλη δουλειά, θα, θα τον είδατε. Είναι πάρα πολύ δραστηριο ε, σε θέματα, 4-5 πήρε και το λόγο, όλη μέρα ήταν παρόν. Από το, το νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι τι 6.30 ήταν παρόν. Οπότε σα διαβεβαιώ ότι ενδιαφέρεται πολύ. Ε, λοιπόν, Δεύτερη ψηφοφορία. Μη στρατιωτικό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GNSS μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου. Καταρχάς θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, πολύ σύντομα θα την κάνουμε αυτή, και μετά μια ψηφοφορία, διότι ψηφίζουμε βάσει της απλουστευμένης διαδικασίας, άρθρο 51. 50.1 χωρίς τροπολογίες και θα είναι ονομαστική ψηφοφορία. Καταρχάς ας δοκιμάσουμε το σύστημα, πώς δουλεύει. Ε, είσαστε έτοιμοι λοιπόν για το Πάσχα είναι η ερώτησή μου. Άρχεται η ψηφοφορία με αυτό το ερώτημα. Πέρας ψηφοφορίας. Βλέπετε τα αποτελέσματα. Δεν βλέπω το αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι είναι έτοιμοι για το Πάσχα. Οι υπόλοιποι θα μείνουν το Πάσχα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα πάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. The is closed. Πέρας. Uh, Δεκτό. 36 υπέρ, 2 κατά, μια αποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η συντομότερη, η συντομότερη ψηφοφορία στην ιστορία μας. Το βλέπω, έχετε επικραθεί, απογοητευτεί, είναι ξεκάθαρο. Α, τι να κάνω, τι να σας κάνω όμως. Now we Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μείωση των εκπομπών για οικονομία και ε, επενδύσεις για χαμηλή κατανάλωση ε, άνθρακος, ETS, που έχουμε μπροστά μας, με άλλα λόγια. Λοιπόν, να σας πω το εξή. Θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ETS είναι σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας στην Ήτρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να αποχωρήσετε την αίθουσα, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε όσο πιο ήσυχα μπορείτε και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα θέλαμε να μείνετε στην αίθουσά μας, αν όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο, σας παρακαλώ να αποχωρήσετε άνευ συζητήσεων δύο φίλοι εκεί στα δεξιά. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Please finished. Now, my goodness. <laughs> okay. Okay. Thank you. Thank you. So, uh... Ευχαριστώ. Το ETS, σημαντικό θέμα για την Επιτροπή Ήτρε, το γνωρίζετε άριστα αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει μια παρουσίαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Γενικό Διευθυντής, ο κ. Ντεμπέκερ θα κάνει την παρουσίαση. Είναι πολύ έμπειρο ε, όσον αφορά τι διαπραγματεύσει και όσον αφορά την πολιτική του κλίματο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντο είναι καθήλυνα αρμόδια, η Ήτρε εμπλέκεται σύμφωνα με το άρθρο 54. Και έχουμε κοινή αρμοδιότητα κυρίως όσον αφορά τα άθρα που αφορούν τη διαρροή άνθρακα πολύ σημαντικό για όλες τις βιομηχανίες πώς ε, να το αντιμετωπίσουν. Πόροι, οικονομική υποστήριξη για τον ενεργειακό τομέα, αποδοτικότητα, εξυγχρονισμός, καινοτομείο, ταμείο καινοτομίας, εξυγχρονισμός, σημαντικότατο θέμα για την Επιτροπή μας. Έχουμε πολλές ευθύνες όσον αφορά το ζήτημα αυτό Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι σημαντικότατη η συζήτηση για μας. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, παρακαλώ προβείτε στα αρχικά σας στεναρτήρια σχολεία σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Με μεγάλη χαρά ξεκινώ τη συζήτηση μαζί σας. Θέλω να ακούσω τι απόψεις σας. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε όσον αφορά την κλιματολογική αλλαγή. Ήταν ιστορική συμφωνία των Παρισίων. Ποιο είναι το ιστορικό της συμφωνίας, δηλαδή ότι όλος ο κόσμος συμμετέχει στην προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το υπογραμμίσουμε ποτέ όσο πρέπει. Όχι μόνο για μας σημαντικό, για τις αναδυόμενες οικονομίες και είπα ακόμα συμμετέχουν στις προσπάθειες αντιμετωπίσεως της αλλαγής του κλίματος. Έχουμε φιλόδοξο στόχο, πολύ πιο κάτω από την αύξηση κατά δύο βαθμούς Κελσίου και αυτό που θα ήθελα να παρουσιάσω για τη σημερινή συζήτηση όπου θα μιλήσουμε βασικά για το ETS, για το εμπόριο ρήπων, ανταλλαγή ρήπων, είναι ότι έχουμε σημαντική κοινοτομία Συμφωνία των Παρισίων, ότι όλες οι χώρες έπρεπε να υποβάλουν σχέδια πολιτικής. Και στα σχέδια αυτά πολιτικής, που είναι καινοφανές αυτό, έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, τι σχεδιάζουν να κάνουν για την ενέργεια, για τις επενδύσεις, για την εξοικονόμηση άνθρακα ε, και για τις μεταφορές και όσον αφορά το εμπόριο ρήπων για τιμολόγηση του άνθρακα και πάνω από τις μισές χώρες του κόσμου σχεδιάζουν να έχουν συστήματα ανταλλαγής ρήπων ή πίστοσης ενεργειακής όπως το ETS. Και στο χάρτη βλέπετε ότι ε, αυτό του είδους το εμπόριο που έχουμε στην Ευρώπη δημιουργείται και στην Κίνα και ο πρόεδρος της Κίνας, ο κ. Τζιζιμπίνγκ, αναγνέρωσε στην σύνοδο το Σεπτέμβριο πέρσι ότι μέχρι το 2017 θα ψηφίσουν την νομοθεσία και το 2020 η κινέζικη, η κινέζικη αγορά θα είναι παρα... διπλάσια της αγοράς άνθρακα της Ευρώπης. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική αλλαγή για τη σημερινή συζήτηση για τη διαρροή του άνθρακα και πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα να συνοψίσω πού βρισκόμαστε. Οι, οι ηγέτες της Ευρώπης, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, κατέληξαν σημαντικό τα συμπεράσματα το 2014, υπολόγισαν το στόχο, είπαν τουλάχιστον 40% μείωση στην εσωτερική, ε, στις εκπομπές εσωτερικές σε σχέση με το 1990 έκανε στάθμιση μεταξύ του ETS που είναι για αυτούς που παράγουν πολλές εκπομπές και την, τον μερισμό των προσπαθειών για εκείνους που εκπέμπουν ε, λιγότερες ποσότητες που είναι στόχος των 100 μελών. Για τον επιμερισμό των προσπαθειών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει πρόταση και πριν το καλοκαίρι φέτος θα την υποβάλει την πρόταση. Αλλά πρέπει να τα δείτε και τα δύο στοιχεία σαν μια δέσμη με τον σαν πακέτο. Έτσι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τον Οκτώβριο 2014 έβλεπαν το όλο θέμα. Λοιπόν, ε, ξέρετε ποιοι είναι οι στόχοι για το ETS 43% βάση του 2005 και αυτό μεταφράζεται σε αιτήσια μήνυση 2,2% και τότε το μερίδιο των ε, δημοπρασιών παραμένει σταθερό 57% και αυτό είναι πολύ σημαντικό πολιτικό στοιχείο στο επίκεντρο, στην καρδιά των αποφάσεων που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Μια άλλη σημαντικότατη πολιτική απόφαση ήταν η εξίσουτα των αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν ότι ένα σύστημα ελεύθερης διανομής για να αντιμετωπιστεί η διαρροή του άνθρακα θα πρέπει να συνεχιστεί σε σύστημα ε, και χωρίς αλλαγή νομοθεσίας ε, το σύστημα θα έλυγε, θα εξέπνεε ε, το 2025. Άρα το θέμα που συζητούμε σήμερα εδώ είναι το πώς θα συνεχιστεί το σύστημα εντός του ορίου που καθορίζεται, κυρίως το μερίδιο των δημοπρασιών του 57%, 43% δηλαδή είναι διαθέσιμο δωρεάν. Λοιπόν, στο επίκεντρο αυτού έχουμε το σύστημα βαθμολόγησης που θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ε, και θα έρθω σε αυτό σε λίγο. Τώρα έχουν δημιουργηθεί και διάφορα ταμεία για να ενθαρρύνουν την καινοτομία, να ενθαρρύνουν τον εξυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα και ιδιαίτερα να επιταχύνουν τον εξυγχρονισμό ε, όσον αφορά τα φτωχότερα κράτη-μέλη που είναι γνωστά σαν κράτη του άθρου 10 γάμα, 10 σύλλα την οικό. Λοιπόν, στη διαρροή άνθρακα πάμε τώρα. Τώρα, το τι μπορούμε να δώσουμε δωρεάν στις εταιρείε είναι κάτι που περιέχεται σε αυτό ε, το τομέα. Έχουμε ένα σύστημα κατά προϊόν βαθμολόγησης, αποτίμησης. Η παραγωγή είναι το τι παράγεται σε ποσότητα και μετά είναι ο παράγων διαρροής άνθρακα. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία τα οποία περιγράφονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει και ενδεχόμενος ε, παράγων συντελεστής διόρθωσης, διορθωτικός συντελεστής. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην ε, πρόταση. Έχουμε εγκάσιο παράγοντα ε, που δεν θα εφαρμοστεί τελικά αυτός ο παράγον που ανέφερα και θέλουμε να λαχιστοποιήσουμε εάν δεν συμβαίνει αυτό ήδη, τον αντίκτυπο που θα έχει ο διορθωτικός αυτός συντελεστής σε όλους τους τομείς. Θα διοργανώσουμε τεχνικό σεμινάριο που θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο, αυτό θα γίνει σύντομα, για να ζητήσουμε από παρατηρητές της αγοράς ποια είναι η άποψή τους. Τι θεωρούν όσον αφορά το μέγεθος, το ύψος που θα έχει αυτός ο διευθυντικός συντελεστής. Πιστεύουμε ότι τελικά ο συντελεστής αυτός θα έχει ε, ε, μικρή, μικρό αντίκτυπο. Ποιο είναι το... Θα έχουμε καλό, καλή προσέγγιση όσον αφορά τους παράγοντες που προανέφερα με αυτή την προσέγγιση, όσον αφορά το σύστημα βαθμολόγησης και τα όρια. Δηλαδή το πόσο μπορεί να εκπέμψει σαν ένα προϊόν, ποσότητα διοξιδίου του άνθρακο σαν ένα προϊόν. Είχε καθοριστεί το 2008. Κάναμε υπολογισμού και προ, προβολέ μέχρι το 2030. Ξέρουμε ότι θα υπάρχουν σημαντικέ τεχνολογικέ εξελίξει. Λοιπόν, πώ αυτέ θα ληφθούν υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ε, εμεί, όπω δείχνουν και οι έρευνε, θα έχουμε κατά μέσο όρο 1% τεχνολογική εξέλιξη που θα οδηγήσει σε αυ, πιο αυ, αυστηρά, αυστηρή βαθμολόγηση και στόχους. Εκείνοι που δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά θα έχουν μισό της εκατό και αυτοί που θα πάνε καλύτερα θα έχουν 1,5% και θα υπάρχει και διαδικασία για να επικυρώνουν τα στοιχεία. Ποια είναι τα ωφέλη της προσεγγίσεως. Εσείς υιοθετείτε την νομοθεσία και όλοι οι βιομηχανικοί φορείς θα γνωρίζουν σε ποια κατηγορία βρίσκονται και θα γνωρίζουν ποια ποσότητα ανακατανομής θα γίνει, θα δημιουργηθεί μια ασφάλεια, μια βεβαιότητα της επιχειρήσης και θα μυθεί η καινοτομία, διότι υπάρχουν κάποιοι που λέγουν ότι κάνουμε μια πρόβα για το σύστημα βαθμολόγησης. Αυτοί που πήγανε πολύ καλά κατά το παρελθόν θα βγουν εκτός. Θα, θα χάσουν τα ωφέλη της καλής απόδοσης τους. Θα πρέπει να επιβραβεύουμε την καινοτομία μέσω καθορισμού της βαθμολόγησης και αυτό προτείνουμε να κάνουμε. Είναι κάτι απλό, είναι προβλέψιμο ε, και αντικατοπτρίζεται στην οδηγία και δεν θα πρέπει να περάσει μέσω επιτροπολογίας. Κατά το παρελθόν πολλά από αυτά αποφασιζόταν μέσω επιτροπολογίας και μέσω καλύτερης θεσπίσεως ε, νομοθεσίας ε, θέλουμε να συμπεριλάβουμε περισσότερα στοιχεία στην οδηγία. Για τη βαθμολόγηση, το σύστημα βαθμολόγησης, το επικαιροποιημένο σύστημα είναι 1% κατά μέσο όρο ε, ενημέρωση των στόχων και της βαθμολόγησης. Γιατί μεταξύ του 2008 και του 2020 και 30 θα δούμε πολλές τεχνολογικές εξελίξεις. Ένα άλλο στοιχείο που λάβαμε υπόψη είναι η καλύτερη ευθυγράμμιση όσον αφορά την αλλαγή της παραγωγής, να συντονιστούμε την αλλαγή της παραγωγής. Πολλοί παραγωγοί έχουν συμμορφωθεί, ε, έχουν πιο σύντομους κύκλους ε, κατανομής η χρονική στέρηση ε, έχει μειωθεί και μπορούμε να έχουμε συμμετρική προσέγγιση. Περισσότερη παραγωγή, λιγότερη παραγωγή, περισσότερη δωρεάν κατανομή, λιγότερη ανάλογα με τον οικονομικό κύκλο. Πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να αποφύγουμε ε, την ε, γραφειοκρατία στο βαθμό του δυνατού, διότι κυκλοφορούν κάποιες προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες εάν αυτές ακολουθηθούν θα δημιουργήσουν μεγάλη αύξηση της γραφειοκρατίας και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και πιο σημαντικό σε επίπεδο των επιχειρήσεων. Προσπαθούμε λοιπόν να περικόψουμε τη γραφειοκρατία και αυτό αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Juncker και γι' αυτό στην νομοθεσία μας έχουμε, ε, προσπαθήσαμε να προστεύσουμε όσο πιο στο βαθμό του δυνατού το σύστημα. Άλλο στοιχείο για την ευθυγράμμιση με την αλλαγή της παραγωγής είναι το απόθεμα για τις νεοεφείς, νεοεσερχόμενες εταιρείες. Αν μια επιχείρηση κάνει μεγάλη επένδυση μπορεί να έχει άλλη προσέγγιση, ξεχωριστή προσέγγιση όσον αφορά την, ε, την άδεια που τις δίνουμε για εκπομπές. Και μετά είναι οι ομάδες που έχουμε στον τομέα της διαρροής άνθρακα. Έχουμε έναν κατάλογο αρκετά μακροσκελή, πάνω από 150 τομείς συμπεριλαμβάνει και στον κατάλογο βλέπει κανείς ποια είναι τα ευάλωτα σημεία τη διαρροή άνθρακα. Βλέπετε αν είσαστε ευάλωτοι στον ανταγωνισμό με τις από τις περιοχές του κόσμου που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Α, αυτό το σύστημα λοιπόν όμως έχει γίνει κάπως ανεξέλεκτο. Μειώσαμε τον αριθμό των τομέων, έχουμε περίπου 50 σημαντικούς ενεργοβόρους τομεί και ξέρουμε ότι 75% των αδειών που χορηγούνται έρχονται από τρει τομεί Από το Χάλιβα, από το τσιμέντο και από τα χημικά. 75% από αυτά παράγονται σήμερα. 50 ενεργοβόροι τομείς. Αυτό είναι μεγάλη απλούστευση. Είναι σημαντική αυτή η απλούστευση ε, και είναι σημαντικό να μην δίνουμε πάρα πολλές άδειες. Ε, έχουμε δύο κατηγορίες όσον αφορά τη ροή του άνθρακα. Εγκαταστάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο, αυτές παίρνουν 100% του συστήματος βαθμολόγησης και μονάδες που είναι χαμηλού κινδύνου που παίρνουν το 30% ε, της βαθμολόγησης. Ποιες είναι χαμηλού κινδύνου, τι σημαίνει χαμηλός κινδύνος. Κάποιες εταιρείες μπορούν στην τιμή των προϊόντων να ενσωματώσουν ένα κομμάτι του κόστους που δημιουργείται από πλευράς ETS, από τον άνθρακα. Και υπάρχει οικονομική τεκμηρίωση εκεί που δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις μπορούν να περάσουν να περάσουν εκεί ένα κομμάτι του κόστους στη δημολόγηση. Πόσο, ποιο ποσοστό του κόστους μπορούν να μετακυλήσουν και εξυπηρετούμε καλά τις μονάδες υψηλού κινδύνου, διότι αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο, δεν θέλουμε να φύγουν βιομηχανίες από την Ευρώπη, κυρίως να μην φύγουν λόγω της πολιτικής μας για τον άνθρακα και για το κλίμα. Θέλουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να κάνουν καινοτομίε, ούτως ώστε αναμονάδα παραγωγής να είναι χαμηλότερες οι εκπομπές. Τώρα, χρειαζόμαστε διορθωτικό συντελεστή. Αν τα πάμε καλά όσον αφορά τον κατάλογο, αν τα πάμε καλά όσον αφορά την παραγωγή και αν τα καταφέρουμε καλά όσον αφορά τη βαθμολόγηση, δεν χρειάζεται ο διορθωτικός συντελεστής και αυτό που ήταν σημαντικό στοιχείο που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει, αυτό το σημαντικό στοιχείο που συζητήσουμε με τη βιομηχανία. Λοιπόν, διαρροή άνθρακα είναι ένα κομμάτι του θέματος. Καλύτερη προστασία όσον αφορά τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, προστασία ανταγωνισμού με εταιρείε που δεν υπόκεινται σε περιορισμού όσον αφορά τον άνθρακα όπω στην Ευρώπη. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τον εξυγχρονισμό Θέλουμε να ενθαρρύνουμε επενδύσεις σε νέες καλύτερε τεχνολογίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τρεις φορεί για να επιτευχθεί αυτό. Και το προτείναμε διότι έτσι πιστεύανε και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Καταρχάς, θέλουμε για τα κάτι μέλη με χαμηλό εισόδημα να έχουν τη δυνατότητα για τον τομέα παραγωγής ενέργειας ίσχυω να δίνονται δωρεάν άδειε. Είναι το άρθρο 10C για εκείνους που θέλουν τις λεπτομέρειες. Δεύτερο ταμείο είναι το Ταμείο για την Καινοτομία. Το Ταμείο για την Καινοτομία ήταν σημαντικότατη μεταβλητή που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν συζητούσαμε το απόθεμα σταθερότητα της αγοράς. Έχει ύψος 450 εκατομμύρια άδειε. Αν πάρετε την τιμή του άνθρακα, αυτή δεν, αυτό είναι πολύ ψηλό, μεταξύ 5 και 10, βλέπετε ότι μιλάμε για ένα ταμείο με πολλά δις ευρώ για την ιδιωτική βιομηχανία, τον ιδιωτικό τομέα, για βιομηχανία που επενδύει σε καινοτομίε για χαμηλή εκπομπή άνθρακα. Αυτό το Ταμείο Καινοτομία σημαντικό το, στοιχείο, σημαντικό ήταν και στι συζητήσει σα, από ό,τι θυμάμαι, για το αποθεματικό για τη σταθερότητα τη αγορά. Εδώ σε αυτή την επιτροπή το συζητήσαμε και χαίρομαι, είμαι περήφανο που αυξήσαμε το ποσοστό και φτάσαμε στα 450 εκατομμύρια ευρώ και μετά έχουμε το Ταμείο Εξυγχρονισμού για χώρες με χαμηλό εισόδημα, όπου χρειάζεται πολύς εξυγχρονισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορεί να ενθαρρυνθεί και είναι το Ταμείο Εξυγχρονισμού λοιπόν, σημαντικότατος φορέας, 310 εκατομμύρια άδειε και πολύ σημαντικό ποσό σε χρήμα αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Ταμείο Καινοτομία, τι έχω να πω. Δεν είναι μόνο θέμα μεγέθους, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσουμε την ενθάρρυνση της καινοτομίας ε, και επενδύσει σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Θα τονίσουμε σε ριζοσπαστικές νέες τεχνολογίες ή στην προσέλκυση επενδύσεων. Στον βιομηχανικό τομέα ίσως να βρουν μια ριζοσπαστική τεχνολογία ε, για να παράγουν ε, προϊόντα με χαμηλότερο εκπομπή ανθράκα όπως είναι στη Χαλιβουργία. Θα επενδύσουμε εκεί ή θα επενδύσουμε σε δίκτυο για ταχεία φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουμε την καινοτομία που ενθαρρύνει τις επενδύσεις ε, εν συγκρίση με χρήση άμεση του Ταμείου για εκείνους που θέλουν να κάνουν επενδύσεις και ρίχνουμε άμεσα τις επενδύσεις. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού είναι για τα κράτη-μέλη που είναι 10 χαμηλού εισοδήματο και αυτό το Ταμείο Εξυγχρονισμού ζητήθηκε κυρίως από τα κράτη-μέλη εκείνα που δεν θα ωφεληθούν από το Ταμείο και θέλουν να δουν να υπάρχει διαφανής διαδικασία σχετικά με την λειτουργία του Ταμείου. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην ε, αρνηθούμε κάτι σε οποιονδήποτε, σε κανένα κατοσμέρος να μην το αρνηθούμε, να έχουμε διαδικασία, να μην υπάρχει βέτο, να υπάρχει θέμα πλειοψηφία και εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή Ταμείο Καινοτομίας. Τρίτο στοιχείο, άρθρο 10C που σας είπα, ε, είναι και πιο σημαντικό σύστημα ενθάρρυνσης που συμπεριελήφθη ε, δωρεάν ε, χορήγηση αδειών σε χώρες φτωχές για τον τομέα παραγωγής ενέργειας να διευκολύνουμε τις επενδύσεις μιλάμε για σημαντικά ποσά οικονομικά δισεκατομμύρια ευρώ άρα είναι πολύ σημαντικό σύμφωνα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε μια ανταγωνιστική διαδικασία που θα σέβεται πλήρως τους κανόνες περικρατικών ενισχύσεων και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σύστημα ανταγωνιστικού ε, συστήματος υποβολής ε, προσφορών που θα είναι μια διαδικασία σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς και διαφανής. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό στα πλαίσια της Ενεργειακής Ενώσεως και στα πλαίσια της της ε, δημιουργίας της ε, ενιαίας αγοράς για τον ηλεκτρισμό. Αυτά είναι τα στοιχεία, ήταν κάπως τεχνικά τα στοιχεία, δεν ήθελα να αναφέρω πολλές λεπτομέρειες, ταυτόχρονα να δώσω επαρκείς λεπτομέρειες για να διευκολύνω τις συζητήσεις. Οι δύο πυλώνες είναι διαρροή άνθρακα, πώς να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εταιρείε στη παγκόσμια αγορά και θετική προσέγγιση να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις στην καινοτομία, επενδύσεις που οδηγούν σε ένα μέλλον με χαμηλή ε, παραγωγή άνθρακα που θέλουμε αυτό είναι το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την και αυτή παρουσίαση. Μας εξηγήσατε πολλά από τα όσα βρίσκονται στο σύστημα. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον δικό μας εισηγητή να μας απαντήσει πώς το αντιμετωπίζει. Ο κύριος Φέντερ λέει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντελπέκε που ήρθε για μια φορά ακόμα στην ε, συνεδρίασή μας για να συζητήσουμε ε, το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις, τους ε, υπαλλήλους. Τελευταία έχω πει πως βλέπω εσάς περισσότερο από την οικογένειά μου και μάλλον αυτό έτσι θα συνεχίσει. Πάντως μέχρι στιγμής έχουμε συναντηθεί με προσώπους 8 κρατών μελών και εκπροσώπους 20 βιομηχανικών κύκλων με ε, ιδρύματα, με πανεπιστήμια, με ερευνητικά κέντρα και με τον κλάδο της ενέργειας. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε το θέμα της ε, διαρροής άνθρακα δεν σήμερα το απόγευμα. Ε, ήμουνα στην... Ε, Πολωνία Υπουργός Ενέργειας και έχω επισκεφθεί και το σχετικό Υπουργείο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε θα συνδυάσουμε εδώ ό,τι ακούσαμε από τα email που λάβαμε, από τους ενδιαφερόμενους, από τις συναντήσεις που κάναμε και η γνωμοδότηση αυτή θα συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή μας 23 Μαΐου. Η τελευταία η προθεσμία υποβολής τροπολογιών θα είναι η τελεία, η, το τέλος Μαΐου με επιθανή ολομέλεια α, μετά το καλοκαίρι. 13 Οκτωβρίου στην Επιτροπή ε, πριν, ε, δύο μήνες δηλαδή πριν την Επιτροπή ε, ΕΜΒ για τους συμβιβασμούς. Ξέρουμε πως σε αυτή τη θητεία με την Ήτρε δεν μπορώ να πω ότι τα έχουμε πάει ε, εξαιρετικά καλά στις ε, ψηφοφορίες μας γιατί χάσαμε κάποιες επιτροπές και στην Ολομήλεια οπότε θα πρέπει αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε εγώ θα προσπαθήσω να πετύχουμε έναν καλό και σταθερό συμβιβασμό και για το λόγο αυτό θέλω να σας παροτρύνω όλους εδώ να ενδιαφερθείτε και να είστε δραστήριοι σε ε, πρώιμη φάση πάντα η πόρτα μου ανοιχτή για τους συναδέλφους από όποιο ε, κόμμα και να προέρχονται. Η Ήτρα είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τόσο επιθυμεί ο κλάδο. Αλλά τελικά αυτό που χρειάζεται είναι η πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Και νομίζω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με, την, με τον εισηγητή, τον κύριο Ντάνκαν στην Επιτροπή ΕΝΒΗ και εγώ πηγαίνω σε όλες τις σκιώδες συναντήσει της ΕΝΒΗ έτσι ώστε και να ακούσω και να ρωτήσω τους ενδιαφερόμενους που παρίστανται σε εκείνες τις συναντήσεις. Τελικά είναι, το βασικό είναι να καταλήξουμε σε μια λογική προσέγγιση η οποία θα ε, φέρει μια ισορροπία μεταξύ των βιομηχανικών και των ε, οικολογικών συμφερόντων. Καταρχήν, λόγω του πολύ ε, επίμονου Προέδρου μας, ε, η θέση μας ε, για το φάκελο αυτό είναι πολύ πιο ισχυρή από ήταν ποτέ στο παρελθόν. Έχουμε αυτή τη στιγμή μοιράσει τις ευθύνε και τις αρμοδιότητες με την ΕΜΒΗ στα πιο σημαντικά θέματα που είναι σημαντικά για τον κλάδο, δηλαδή την διαρροή, την δωρεάν κατανομή αδειών κτλ. Ή για να το πω και πιο απλά στο ΤΕΝΣΥ. Στα στοιχεία αυτά θα αναφερθώ κατά τη διάρκεια τη σύντομη παρουσίας που θα κάνω και θα είναι και στη βάση τη γνωμοδότησή μου, παρόλο που υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να δούμε. Καταρχήν, ε, τα μέτρα για την ελεύθερη κατανομή και για τη διαρροή άνθρωπων. Εδώ θέλουμε ένα οικονομικά αποδοτικό σύστημα μείωση εκπομπών που θα μα διατηρήσει ανταγωνιστικού για όσα ευρωπαϊκά συμφέροντα αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα από την παγκόσμια αγορά. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεται αυτή η δημοπρασία των αδειών, αλλά για κάποιους κλάδους βιομηχανικούς θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ε, ελεύθερη δωρεάν αυτή η κατανομή ως εξαίρεση προς το γενικό κανόνα, έτσι ώστε να αποφύγουμε τη διαρροή άθρακα. Τι βλέπω τώρα πως υπάρχει ένας καθορισμένος αριθμός αδειών σύμφωνα και με την πρόταση της Κομισιόν και αυτές δεν είναι αρκετές έτσι ώστε να μοιραστούν σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μερικές δύσκολες επιλογές στην Επιτροπή μας. Τα διαφορετικά στοιχεία της ελεύθερης κατανομής συνδέονται άμεσα και θέλω να κάνω ένα πακέτο, πρόταση πακέτο για τα θέματα στο οποία επηρεάζει η ΙΤΡΕ. Θέλω η καλύτερη αποδοσή να ε, ευνοείται Άρα δηλαδή ένα σύστημα δωρεάν κατανομής που θα ελαχιστοποιεί ε, που θα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο να επιβάλλουμε το συντελεστή της ε, διακλαδικής ε, επίδρασης. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε αν είσαι ο πιο ποδοτικός στην κατηγορία σου ή ο λιγότερο ποδοτικός. Και θα πρέπει οι κανόνε εκεί να είναι ρεαλιστικές, να αποτελούν ένα στοιχείο που θα μας ενθαρρύνει να τα πάνε καλύτερα στο μέλλον. Περισσότερο δε οι κλάδοι οι οποίοι ε, εγκυμονούν τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Και δεν μπορούμε εμείς εδώ να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι και υπέρ των δέων περίπλοκο. Το Ταμείο Καινοτομία. Εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να έχουμε καινοτομίε στην τεχνολογία για τη μείωση των εκπομπών, να είναι ένα, ένα όχημα ανάπτυξης αυτών των τεχνικών που θα πρέπει να συμπεριλάβουν και χαμηλές εκπομπής άνθρακας καινοτομίε στο βιομηχανικό κλάδο και θα πρέπει να δούμε και τα ορόσημα τα οποία θα τοποθετήσουμε έτσι ώστε να αξιολογείται η πρόοδος. Τώρα για τις βαθιές μειώσεις που έχουμε στα πλαίσια της μακροπρόθεσης νοτατριγικής το 80 με 95% των εκπομπών μέχρι το 2050 χρειαζόμαστε ένα ταμείο με περισσότερα κονδύλια έτσι ώστε να μοχλευθούν με τα ιδιωτικά για να έχουμε πραγματικά τεχνολογία εκμή στον κλάδο και θα πρέπει το ταμείο αυτό να μην είναι πολύ περιπλοκό στη χρήση του και θα πρέπει η βιομηχανία να μπορεί να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα κονδύλια. Τρίτον, ο εξυγχρονισμό και το Ταμείο Εξυγχρονισμού είναι το 10C. Για παράδειγμα, εδώ στο Ταμείο αυτό για τη μεταβατική δωρεάν κατανομή για τον εξυγχρονισμό του κλάδου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την επανεπένδυση στον εξυγχρονισμό του κλάδου τη ενέργεια στα 10 ε, ε, χαμηλοτερου εισοδηματο εισοδήματος κράτη-μέλη. Δηλαδή, μακροπρόθεσμοι στόχη για το κλίμα και σεβασμό των εθνικών προαιρετήτων σε ε, παραλληλισμό. Τώρα, και θα το κλείσω εδώ κύριε Πρόεδρε, για τον εξυγχρο... το Ταμείο Εξυγχρονισμού χρειαζόμαστε να εξεύρουμε την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ε, ρόλων, έτσι ώστε να δούμε πώς η ΕΤΕ, τα κράτη-μέλη δικαιούχοι, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή θα συνδυάσουν τις προσπαθειές τους. Και το τελευταίο που έχω να πω αυτή τη στιγμή συνεχίζει τη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την μετά το Παρίσι εποχή. Είναι πολύ σημαντικό κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό. Θα μπορείτε να πείτε και δύο λόγια στο τέλος. Ναι, Οπότε για την Συμφωνία των Παρισίων θα επανέλθω αργότερα γιατί θα, και θα κρατήσω την ανάσα μου μέχρι να μου δώσετε ξανά το λόγο. Ναι, μετά τη συζήτηση. Μετά τη συζήτηση έχουμε πάλι σοβαρά θέματα. Φαντάζομαι που ο συνάδελφος, ο από την Επιτροπή ΕΝΒΗ, ο Ιαν Ντάνκαν, θα ήταν εδώ μαζί μας. Αυτό φανταζόμουν, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε συνεχή επαφή με τους βασικούς είδες, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει. Ναι. Ίσως όμως οι συνάδελφοί του Μήπως κάποιοι από την ECR θα μπορούσαν να τον πείθουν να έρχονται εδώ για τα πιο σοβαρά θέματα που έχουμε στο τραπέζι. Τώρα, πολιτικές ομάδες, ΕΛΚΑ. Η κυρία Ντελάγκη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ακούσω το Φρέντερικ τώρα για την κατάσταση μετά το Παρίσι. Τον κόψατε και πραγματικά μας έχετε σε μεγάλη αγωνία τώρα. Γιατί ε, ε, θέλαμε μια συνολική ε, γενική συζήτηση πριν μπούμε στις τεχνικές λεπτομέρειες και στη δική μας Επιτροπή εδώ αλλά και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό είναι από τα πρώτα ζητήματα. Τι θα κάνουμε τώρα μετά το Παρίσι. Και πρέπει να απαντηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φρέντρικ και τους συνεργάτες του γιατί έκανα πολλές συνεδριάσεις με τους ενδιαφερομένους και τους κοιόδης ηγητές. Ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εμείς το ETS το βλέπουμε βεβαίως σημαντικό και θέμα ευθύνης για τον πλανήτη και τις επόμενες γενιές, αλλά είναι και πάρα πολύ στρατηγική σημασίας ε, στη θητεία μας από τα σημαντικότερα ίσως. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το σύστημα εμπορίας εκπομπών και πώς ε, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παγκόσμιο στερέωμα. Χαίρομαι που ορισμένοι τομείς και τους αναφέρετε είναι ε, αναγνωρισμένο ότι εκπέμπουν περισσότερο, αλλά δεν μπορούμε εμείς να είμαστε δύο και τρεις φορές πιο καθαροί από ότι η Κίνα γιατί σηκώνεται και φεύγει η παραγωγή. Και εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να αποβούν και μοιραίε και ανήτικε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και θα χάσουμε στρατηγικά σημαντικούς τομείς, όπως είναι ο Χάλιβα. εγώ θα αναφέρω και τα λοιπάσματα. Το γεγονός ότι αυξάνεται η εξάρτησή μας για αυτούς τους στρατηγικούς τομείς από άλλα μέρη του κόσμου θα ήταν λάθος και σημείωσα όσα είπατε κύριε Ντελμπέκε για τις εξελίξεις στην Κίνα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε χάσει ακόμα τη βιομηχανία μας και δεν είναι μόνο θέμα ETS, είναι θέμα και ανταγωνισμού, αλλά έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να μην σηκωθούν να φύγουν πριν αρχίσουμε εμείς να κινητοποιούμαστε ή άλλες περιοχές του κόσμου. Στη δική μας λοιπόν επιτροπή εναπόκειται Βεβαίως να σεβαστούμε την προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών, αλλά ταυτόχρονα, λέω, η Επιτροπή μας θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη θέση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Είμαστε Επιτροπή Βιομηχανίας στο κάτω-κάτω. Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περισσότερες δωρεάν ε, ε, ε κατανομές σε ορισμένες περιπτώσεις και περισσότερο συντονισμός για να ε, αντιμετωπίζουμε ρεαλιστικά την κατάσταση και την παραγωγή με βάση πραγματικά στοιχεία. Αυτό το καιρό βολιδοσκοπούμε τις διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν και τις επιλογές για να δούμε ποια θα ήταν η πιο ευφύης πρόταση και πιο αποτελεσματική. Πάντως για μας ε, το Λαϊκό Κόμμα τα σημαντικότερα είναι τα εξή. Βεβαίως θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ε, κλιματικής αλλαγής, ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας παγκοσμίω, να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο ε, της λεγόμενης διαρροής άνθρακα, δηλαδή να σηκωθούν να φύγουν οι βιομηχανίες που παράγουν πολύ διοξίδιο και είναι ενεργοβόρες και για την καινοτομία δεν έχουμε δώσει αρκετή προσοχή. Τελειώνω. Ιδιαίτερα μιλώ και δεδομένη τη δική μα αρμοδιότητα και του πεδίου που απασχολεί την Επιτροπή Βιομηχανία. Συγκεκριμένη ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν και κάποιοι τομείς εκτό ETS και επίκειται πρόταση και υπάρχει μια πίεση να συμπεριληφθούν και άλλοι κλάδοι που μέχρι τώρα δεν ε, περιλαμβανόντουσαν και έχουμε κάποιο χώρο στο ETS. Πώς το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρακαλούσα όσοι μιλάτε εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων αν υπερβαίνετε το τρίλεπτο δεν θα μας στάσει ο χρόνος. Ο κύριος ε, Μαχτά παρακαλώ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Πρόεδρε, ε, κάθε φορά που είναι η σειρά μου θα νομίζω ότι έχετε τίποτα προσωπικό. Μου δίνετε το λόγο και υπενθυμίζοντας το χρόνο κάθε φορά. Ε, 17 λεπτά τονίζω μίλησε ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής ναι. Επιτροπής. Δεν θα μιλήσω εγώ 17 λεπτά, αλλά θα προσπαθήσω να πω αυτά που έχω να πω. Και ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική συζήτηση. Άκουσα με προσοχή τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι το σύστημά μας δεν το εφαρμόζει πάρα πολλοί κόσμο <laughs> στην Ιφίλιο. Έτσι. Και εγώ είμαι σαν τον άπιστο Θωμά. Πρέπει να το πιάσω για να το πιστέψω κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνη της στον κόσμο και ποια είναι η πραγματική ιδέα. Πώς ε, όλοι οι φορείς θα έχουν ίση μεταχείριση ή θα υπάρχουν ίση κανόνες παιχνιδιού. Σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τα εργοστάσια. Ε, κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες ε, διαπιστώσεις. Το ETS βεβαίω σήμερα είναι αξιόπιστο για να περιορίσει τι εκπομπέ ρήπων και καλά κάνει. Αλλά θα πρέπει να δούμε ε, τι εξαιρείται. Οι μεταφορέ, η γεωργία, όλα τα μη βιομηχανικά, τι θα κάνουν αυτοί για να μειώσουν τι εκπομπέ ε, των αερίων του θερμοκηπίου. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να έχει ένα κόστος το διεξίδιο του άνθρακα για να ε, καθοδηγηθούν κάπου οι επενδύσεις, αλλά το τελευταίο διάστημα δεν έγινε αυτό. Βλέπουμε πόσο κοστίζει ο τόνος διοξιδίου του άνθρακα, φλετάρει ανισχυτικά με τα 5 ευρώ. Ε, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό. Και ε, υπάρχει και ε, το απόθεμα σταθερότητας για το 2019, αλλά τίποτα ε, δεν μας κάνει να πιστεύουμε ότι μέχρι το 2030 θα έχει φτάσει τα 25 ευρώ. Άρα αυτό δεν είναι παρκές κίνητρο, επαναλαμβάνω, για να φύγουμε από την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Σας ερωτώ λοιπόν, τι γίνεται. Ε, πέρα από το απόθεμα αυτό, το αποθεματικό, έχετε σκεφτεί μια κατώτατη τιμή του τόνου διοξιδίου του άνθρακα. Ε, η Γαλλία έχει κάνει μια πρόταση ε, Corridor Carbon, πώς τη βλέπετε. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Υπήρξε μια πρόταση, δεν μπορούμε να πούμε ότι έλαμψε με την επιτυχία που τη συνόδευσε. Βέβαια δεν έχουν φύγει ακόμα όλες οι επιχειρήσεις, αλλά ούτε και έχουν επενδύσει. Αν δούμε τους κλάδους που μας ενδιαφέρουν, εκείνοι που λέγουν ότι μείωσαν την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, το έκαναν επειδή έκλεισαν τα εργοστάσια, όχι επειδή τα βελτίωσαν ή τα εξυγχρόνισαν για να μειωθούν οι εκπομπές. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, πώς να επανέλθουν οι επενδύσεις. Εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή για τον τρόπο που διαχειρίζονται ε, τις ποσοστώσεις και τις πουλούν τα κράτη-μέλη. Και δεν θα πρέπει να έχουμε απλώς ε, ε, οικονομικά και χρηματικά κριτήρια. Ο στόχος πρέπει να είναι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Θέλω να πω το εξής και με γνωρίζουν πολλοί εδώ και συμφωνούν. Αυτή η μεταρρύθμιση ETS, ξέρω ετοιμάζει το πρόεδρος να με κόψει, δύο δεύτερα παρακαλώ, είναι ε, ένα τεράστιο κατασκεύασμα δυσλειτουργικό και είναι κρίμα γιατί ε, όταν θέλουμε να ε, μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου φτιάξουμε ένα τέτοιο τεράστιο κατασκεύασμα βαρύ και δυσλειτουργικό. Και στα σύνορα θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή και υπολογισμό για το διοξίδιο του άνθρακα και τελειώνω. Τελειώνω. Θέλουμε και ένα ταμείο μετάβαση για τις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο γιατί υπάρχει και κοινωνικό αντίκτυπος. Ο κύριο Φόξ, εξ ονόματο των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρου του συναδέλφου του Χάν Όλαφ Χάνκελ, που δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα να σας διαβάσω την ομιλία του. E το σύστημα το ευρωπαϊκό, το ETS, δεν αρκεί για την καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο και την αύξηση της δημοκρασίας. Για να μειώσουμε τι εκπομπέ. Ε, δεν ξέρουμε αν είναι αποτελεσματικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε τι εκπομπέ τη, αλλά το ποσοστό εισαγωμένων εκπομπών αυξήθηκε εν μέρη λόγω διαρροή άνθρακα και παγκόσμια μετακίνηση των εκπομπών προς Ανατολά. Η αλλαγή του κλίματος είναι παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο απαιτεί μια παγκόσμια λύση. Μια, ένα ευρωπαϊκό σύστημα συνεπώς δεν αρκεί, διότι αγνοεί την παγκόσμια πτυχή της αλλαγής του κλίματος και δημιουργεί ένα παράδοξο οι εταιρείε οι οποίε εκπέμπουν περισσότερο παίρνουν τι περισσότερε εξαιρέσει για να αποφύγουν τον κίνδυνο διαρροή άνθρακα και να βρεθούν σε μειονεκτική ανταγωνιστικά θέση. Όμω το ETS εξακολουθεί να είναι το καλύτερο εργαλείο με βάση την αγορά που έχουμε στη διάθεσή μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπώ θα πρέπει να ηγηθεί μέσω παραδείγματο, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσει τελικά να συνδέσει την αγορά ε, άνθρακό τη με άλλε. Να ενταχθεί το σύστημα με την Ελβετία, την Κίνα, την Αυστραλία ε, και άλλα συστήματα είναι κάτι που συζητείτε. Το επιτυχές αποτέλεσμα σίγουρα θα δημιουργήσει μια ε, ορμή και θα εμβαθύνει τη συνεργασία των αγορών σε διεθνέ επίπεδο. Για να λειτουργήσει το ETS, η δίποτε δημόσια παρέμβαση πρέπει να είναι περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτό θα, θα έχει θετικό αντίκτυπο στι τιμέ. Ευπρόσδεκτο αυτό, διότι η τιμή του άνθρακα σημερινή είναι πολύ χαμηλή. Παρόλο που είχε ανάγκη να περιοριστεί ο αριθμό των τομέων όσον αφορά τον κατάλογο διαρροή άνθρακα και να καλυφθούν οι σημαντικότεροι τομεί, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ταυτόχρονα μεταξύ του περιορισμού αυτού και τη προστασία των ανάντι και κατάντι τομέων που επίση έμεσα επηρεάζονται. Αυτοί οι τομεί πολύ συχνά είναι αποδοτικότεροι από του ανταγωνιστέ στον κόσμο και η παραγωγή του αερίου είναι κάτι που έχει νόημα όσον αφορά το περιβάλλον Τώρα, όσον αφορά το Ταμείο Καινοτομία, να σημειωθεί ότι εταιρείε του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερε, ε, δεν έχουν έλλειψη πόρων για την καινοτομία. Όμω, η επενδυτική του προτεραιότητα ίσω να μην είναι η καινοτομία για τα οικολογικά θέματα. Το Ταμείο θα πρέπει να υπεριστεί σε καινοτομίε όσον αφορά το περιβάλλον, για να αναβαθμιστούν αυτοί οι τομεί και να δημιουργηθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Επίτροπο Μέντα ήδη έχει προβάλει την ιδέα να υπάρξει ένα Συμβούλιο Ευρωπαϊκό Καινοτομία. Εάν δημιουργηθεί αυτό το Συμβούλιο, το ερώτημα είναι πώς αυτοί οι δύο φορείς θα συσχετιστούν εντός του ευρυτέρου θεματολογίου καινοτομία του Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόεδρε. Αυτά είναι τα σχόλια του κύριου Χένκελ. Αν επιτρέπετε να προσθέσω και ένα δικό μου σχόλιο. Ακούσαμε σήμερα το σύστημα βαθμολόγησης, benchmarking, που θα υποθέσει βελτίωση 1% βελτίωση κάθε χρόνο και πάντα. Τι θα γίνει όμως με τις κάπως λιγότερο ανταγωνιστικές ε, βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που όμως είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από τους ανταγωνιστές τους στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Και φοβούμε ότι αυτό που θα κάναμε θα βγάλουμε εκτός αγοράς το λιγότερο αποδοτικό 25% της Ευρώπης, η, η οδήποτε τομέα, χάλιβα, ε, δηληστήρια, τσιμέντο κλπ. Ποιο είναι το καθαρό αποτέλεσμα, η λιγότερο αποδοτική βιομηχανία της Ευρώπης είναι πιο αποδοτική από τους ανταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό θα έχει αποτέλεσμα διαρροή άνθρακα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έριξον, από πλευράς των Προσύνων. Thank Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς δεν λειτουργήσε το ETS ε με τον τρόπο με τον οποίο είχε σχεδιαστεί και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκπομπές ε, άνθρακα μειώθηκαν λόγω οικονομικής κρίσης και όχι λόγω ETS. Πολύ συχνά ε, κοιτάω το σύστημα και διαπιστώνω ότι είναι πολλά τα σημεία στα οποία έχει αποτύχει και δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα για τη μετάβαση προς την ε, χαμηλών εκπομπών ε, παραγωγή και νομίζω ότι σε πολλές φορές ε, στρέφουμε και προς την αντίθετη κατεύθυνση τους παραγωγούς. Καταρχήν, δωρεάν κατανομή. Κάποιες εταιρείες λαμβάνουν περισσότερες άδειε από ό,τι χρησιμοποιούν, από ό,τι χρειάζονται, γιατί η παραγωγή τους είναι χαμηλότερη από τις άδειε τις οποίες έχουν κατανεμηθεί. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να βλέπουμε τα πραγματικά στοιχεία παραγωγής και τον πραγματικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα και να μην έχουμε αυτό το πολύ απέδευτο σύστημα. Και να ακολουθήσουμε μια κλιμακωτή προσέγγιση ε, έτσι όπως γίνεται στη Βρετανία. Δεύτερον, τα έμεσα κόστη του άνθρακα ε, αποτελούν πρόβλημα κατά τη γνώμη μου γιατί ένα σύστημα στο οποίο τα κράτη-μέλη μπορούν να αποζημιωθούν για υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι λογικό. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέγει τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και η βιομηχανία θα πρέπει να επιλέγει αν θα αγοράζει από καθαρό παραγωγό ή από παραγωγό που μολύνει. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή τιμέ αγορά ε, εξαρτώνται από την προσφορά και από τη ζήτηση, όχι τόσο πολύ από το κόστος. Και αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό γιατί κάποιες εταιρείες λαμβάνουν αποζημιώσεις ε, βασιζόμενες σε εσφαλμένους υπολογισμούς και πολλές φορές τελικά όσοι χρειάζονται δεν λαμβάνουν αυτή την αποζημίωση ενώ αντίθετα αυτοί που δεν τη χρειάζονται λαμβάνουν γιατί ζουν σε μια χώρα η οποία ευημερεί περισσότερο και μπορούν λοιπόν να πληρωθούν αυτές τις αποζημιώσεις. Δυστυχώς, και αυτό είναι το τρίτο σημείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί τη λογική πως όλοι θα πρέπει να αποζημιώνονται ε, με επιχειρηματολογία είναι εξαιρετικά ε, πτωχή. Τώρα το τρίτο σημείο είναι η μετάβαση προς τον εξυγχρονισμό του κλάδου. Οι περισσότεροι πόροι από το τρέχον σύστημα ε, προέρχονται από το άρθρο 10C, 10Γ που επιτρέπει Εντάξει, στα κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη βλέπουμε δωρεάν κατανομές έτσι ώστε να έχουμε καθαρότερη παραγωγή ενέργειας. Νομίζω πως αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί στέλνουμε κίνητρα για να διατηρηθούν τον άνθρακα και κυρίως μιλάω για την Πολωνία και άλλες χώρες ή ε, εγκαταστάσεις παραγωγής. Ο κύριος Σιλικιώτης παρακαλώ την ΚΟΕ. Στον Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους μας ε, η ανάγκη για αλλαγή του συστήματος ETS. Όμω η αναθεώρηση του συστήματο εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, όπω αυτή προτείνεται από την Κομισιόν, αντί να έχει ω πρωταρχικό στόχο τη μείωση των εκπομπών, επιδιώκει δυστυχώ την αύξηση τη ανταγωνιστικότητα τη Ένωση και την παροχή δωρεά δικαιωμάτων σε βιομηχανίε που προγραμματίζουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγουν τα τέλη ρήπαση. Εμεί ω ΓΚΟΕΝΤΖΙΕ δεν θέλουμε ένα σύστημα που να ευνοεί τις μεγάλες πολυεθνικές και τα μονοπόλια για να αυξάνουν την κερδοφορία. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι και η κύριοι υπέτειοι των κλιματικών λαών. Επίσης δεν θα στηρίξουμε αλλαγές που ωφελούν τις ανεπτυγμένες χώρες σε βάρος των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Αντιθέτω, θεωρούμε πω η αναβάθμιση των δικτών αναφορά και όποιο εξυγχρονισμό του συστήματο θα πρέπει να έχει πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντο και την ενίσχυση τη ποιότητα ζωή των ανθρώπων. Εξίσου σημαντικό είναι να λαμβάνει υπόψη τι ιδιαιτερότητε των κρατών και δει τι ιδιαίτερε συνθήκε που επικρατούν στα κράτη του Νότου εν μέσω μια φοβερή οικονομική κρίση, εν μέσω μια αδιέξοδη ε, ύφεση στην οικονομία ε, και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Ε, Προ αυτή την κατεύθυνση επίση θα πρέπει να υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα για του μεγαλύτερου ρηπαντέ Επίση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ξέρουν από το σύστημα του μικρού δερματές, εκείνου που δεν επηρεάζουν ε, σοβαρά το ζήτημα και έτσι ε, προστατεύουν ιδιαίτερα ε, μικρές μικρές επιχειρήσεις κυρίως οικογενειακά. Όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει, δεν πρέπει να υπάρξει συναρμόνιση, καθώ σε τέτοια περίπτωση δεν θα αναβάλλονται υπόψη οι ιδιαιτερότητε κάθε χώρα. Δεν πρέπει να υπάρχει κρατική ενίσχυση να είναι η δικαίωμα του κράτου, λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαιτερότητε που υπάρχουν σε κάθε κράτο μέλο. Αντί λοιπόν στόχο να είναι η ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα και η στήριξη των μεγάλων πολυεθνικών, η μεταρρύθμιση του συστήματο λαμβάνω θα πρέπει να προωθεί και νετόμε αλλαγέ με στόχο τα συμφέροντα και τι ανάγκε τη οικονομία, που να βοηθά και στον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση τη κοινωνία, αλλά πόροτα και κύρια στην ποιότητα ζωή των ανθρώπων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Εξ ονόματος της ΕΝΕΦ, e η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης εργάστηκε πάρα πολύ επικοδομητικά και με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό, μας ενημέρωσε με σεμινάρια, και όλους τους ενεχόμενους ε, και τους και για να γίνει μια συζήτηση επί της ουσίας και κοντά στην πράξη και όχι θεωρητική, για να μπορούμε να εργαστούμε και στο μέλλον έτσι, με μέθοδο. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αφορά μόνο το σύστημα εμπορίας εκπομπών, έχει επιπτώσεις και σε πολλά θέματα όπως αυτά που συζητήσαμε χθες για την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και άλλα πολλά και βέβαια γράφεται σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Υπάρχουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες που συζητήσαμε και χθες. Υπάρχει διεθνής ανταγωνισμός και μας είπε χθες ο Επίτροπος Κατάινεν ότι ε, στις νέες ε, συμφωνίες και σε νέα εμπορικά μέσα ε, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του dumping, ε, ιδιαίτερα στη χαλιβουργία. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσουμε και το σύστημα ETS. Δεν είναι μόνο αυτό που αυξάνει το κόστος, αλλά και το υψηλό κόστος στην Ευρώπη και της ενέργειας και της εργασίας. Αν μιλούμε για 20% επαναβιομηχάνηση μέχρι το 2020, πρέπει να τα λέμε και αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, η Κίνα του χρόνου θα εισαγάγει ένα τέτοιο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Το συζητήσαμε και αυτό και αν δείτε ε, ε για τις ε, μολύνσεις και τη ρήπανση από το 2012-2030 θα ε, φτάσουμε εμείς στο 5% και η Κίνα ε, πάνω από 20% και ε, οι αναδυόμενες οικονομίες τώρα είναι στο 43% της ρήπανσης και προσεχώς στο 52% για να δούμε και ποιος θέει. Και το είπε πολύ σωστά σήμερα ο Γενικός Διευθυντής. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δείκτηση, αυτό το benchmarking, η βαθμολόγηση, ε, για να βεβαιωθούμε ότι η δωρεάν ε, παροχή ή παροχή μάλλον δωρεάν δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να πλήττει την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων ε, βιομηχανιών. Θα πρέπει οι πρωτοπόροι να επιβραβεύονται και να μειώνεται και η γραφειοκρατία και σε επίπεδο κρατών μελών ε, και σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο γίνεται. Ε, ακούσαμε και για διάφορα ταμεία, πολύ σημαντικά και το Ταμείο Καινοτομίας και το Ταμείο Εξυγχρονισμού το Ταμείο Καινοτομίας φυσικά για τις επιχειρήσεις είναι ένα κίνητρο για να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες, για να ε, πούμε ότι θα έχει και μεγάλη σημασία το Συμβούλιο Καινοτομίας και το Ταμείο Ξυγχρονισμού είναι υπέρ των 10 κρατών που έχουν χαμηλό εισόδημα και μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει και προστασία του ανταγωνισμού, αντίστοιχη διαδικασία για να λειτουργούν σωστά όλα αυτά τα πράγματα. Very much, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Έχω στον κατάλογο άλλους 11 παρακαλώ συναδέλφους. Για τους σκιώδεις είχαμε πάνω από 3 λεπτά, 3,5 περίπου, κάτι τέτοιο. Για τους υπολείπους συναδέλφους παρακαλώ να μην υπερβείτε το δίλεπτο, διότι δεν θα προλάβουμε με 11 ομιλητές. Πού να τους χωρέσουμε. Κύριε Ζουρούβιχ, πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω η παρουσίαση μας έδειξε ότι έχετε πολύ μεγάλες προθέσεις και επίβολες Να δούμε τι θα γίνει με τη μελέτη αντικτύπου όμως σε αυτό το τομέα διότι από τη μια έχουμε ένα στόχο 20% περισσότερη παραγωγή στην Ευρώπη μέχρι το 2020, επαναβιομηχάνηση, τώρα είμαστε στο 15% με πτωτικές τάσεις. Έχουμε χάσει 8% της παραγωγής από το 2008. Άρα πώς μπορούμε εμείς την παραγωγή στο μέλλον να την ε, προστατεύσουμε με αηφορία και να την προσελκύσουμε και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ο προσωπικός μου στόχος θα ήταν να έχουμε και στόχο για το 2030 για τη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη και προσωπικά θα έλεγα 30% μέχρι το 2030. Εγώ είμαι από την Άνω Αυστρία που έχουμε παραγωγή αυτή τη στιγμή 32%. Νομίζω για τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη αυτό θα έχει τεράστια σημασία. Να δούμε τη μελέτη αντικτύπου που δημιουργούνται οι νέες καλές ποιοτικές θέσεις εργασίας με αηφόρο και βιώσιμη παραγωγή και που μπορεί πραγματικά η Ευρώπη να είναι ηγετική στην παραγωγή των προϊόντων. Δηλαδή από τη μια μελέτη επιπτώσεων, από την άλλη και ένα τεστ μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει πολύ σημασία και πολύ μεγάλη διότι σε αυτές τις νέες τεχνολογίες δραστηριοποιούνται πολλές μικρομεσαίες, δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας και είναι σημαντικό να ελέγξουμε και το κόστος της γραφειοκρατίας όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές αλλά και σε εθνικό. Τι σημαίνουν αυτές οι ρυθμίσεις, τι κόστος θα μας έρθει, πώς το υπολογίζουμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντελμπέκε που πραγματικά κάνει προσπάθειες να αποτρέψει το γραφειοκρατικό άχθος για τις επιχειρήσεις και να είναι γίνεται πιο διαφανής ρυθμίσεις. Άλλο σημαντικό όμως για τη μείωση ε, του διοξιδίου του άνθρακα ε, έχει να κάνει και με τις εισαγωγές. Εισάγουμε 400 δισεκατομμύρια τώρα ενέργεια, ε, ε, ορυκτά καύσιμα δηλαδή. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Ε, μερικές προτάσεις μόνο για την έκθεση ε, εν ώψη της εκπόνησης. Ε, σε ό,τι αφορά το έμεσο κόστος για τομεί ε, που φεύγουν από την Ευρώπη λόγω διοξιδίου του άνθρακα. Υπάρχει πρόβλεψη για αποζημίωση από την Ευρώπη, για το έμεσο κόστος, ιδιαίτερα για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή δεν θα πρέπει να μετακυλίεται στο κόστος αυτό στον τελικό καταναλωτή, αλλά θα πρέπει από τα δικαιώματα ε, των δημοσπρασιών να καταβάλλεται αυτό το κόστος. Επίσης για την κοινοτομία θα πρέπει να έχουμε υπόψη όλες τις νέες τεχνολογίες για χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Ε, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην έρευνα και σε προϊόντα καινοτόμα, πρωτοπόρα ε, της έρευνας που μειώνουν αποδεδειγμένα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την παραγωγή αερίων δηλαδή, θερμοκηπίου και θα αποδώσουν σε μέσω πρόθεσμη βάση και θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε ε, τα εφή δίκτυα, τις ευφύης ε, πόλης ε, κτλ. Και επίσης δεν θα πρέπει να μειωθεί το ποσοστό των δικαιωμάτων από το 57% όπως έχει καθοριστεί με τρόπο σταθερό στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρινς. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, διαβάζοντας όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερη δυσκολία γιατί δεν βλέπω αυτό το οποίο εγώ θα ονόμαζα μια πραγματική επιπτωσιολογική μελέτη για το τι θα δημιουργήσουμε ε, και πώς αυτό θα επηρεάσει τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Βεβαίως πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές θερμοκηπίου σε όλο τον πλανήτη και τονίζω σε όλο τον πλανήτη. Πώς λοιπόν επηρεάζουμε και τι στοιχεία έχουμε και πώς θα έχετε αναλύσει τα δεδομένα αυτά από την πρότασή σας για το τι θα σημαίνει αυτό σε αριθμό θέσεων απασχόλησης. Και δεύτερον, ε, απώλεια ε, επενδύσεων. Να μιλήσουμε για διαρροή επενδύσεων. Μιλάω για μια εταιρεία η οποία δεν φεύγει από την Ευρώπη, αλλά επενδύει εκτός Ευρώπης, ε, δεν αναπτύσσεται δηλαδή εντός της Ευρώπης. Άρα λοιπόν είναι μια απώλεια ευκαιρίας, επενδυτικής ευκαιρίας ή αναπτυξιακής ευκαιρίας. Επίσης, αν ε, είναι κανείς ε, σαν τη Λετωνία για παράδειγμα, που είναι πολύ πράσινη χώρα. Δεν είμαστε στο 50% των εκπομπών ε, του ETS που είναι η υπόλοιπη Ευρώπη, είμαστε στο 22%. Αυτές λοιπόν οι εκπομπές που προκύπτουν επειδή ακριβώς είμαστε τόσο πράσινοι θα αποζημιωθούν έτσι ώστε η βιομηχανία μας να μείνει στη χώρα. Γιατί Εάν κανείς αποκομίζει κέρδος από την πώληση εκπομπών, δυνατοτήτων εκπομπών, τότε θα έπρεπε τα έσοδα αυτά να χρησιμοποιηθούν για να επενδυθούν σε κάποιο άλλο κλάδο ο οποίο έχει εκπομπέ ενέργεια, στις για παράδειγμα. Άρα λοιπόν το σύστημα το οποίο στείλουμε είναι σωστό, ενώ αν μπορούν κάπου να γίνει εξοικονόμηση από τις εκπομπές, από ε, το ποσοστό εκπομπών, μήπως θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά με έναν άλλο τρόπο για να σώσουμε θέσει απασχόληση που πράγματι χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν να δούμε ποια είναι η πραγματική επιπτωσιολογική μελέτη για τις α, θέσεις εργασίας. Η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ κύριε ε, γιατί πρέπει να τα καταφέρουμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούσουμε τους εμπλεκόμενους. Είναι οι χρειές, είναι η στόχευση. Και καλωσορίζω αυτή την πολύ σφαιρική προσέγγιση του Φρέντερικ που ακούει όλους και όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται εδώ για μάχη μεταξύ των βιομηχανιών και του περιβάλλοντος. Όχι, έχει να κάνει με το βιώσιμο μέλλον που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για τις επόμενες γενιές, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα στις βιομηχανίες μας. Θα πρέπει να τα καταφέρουμε και στα δύο επίπεδα. Τώρα, για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και για το πώς χρησιμοποιείται ε, οι χρησιμοποιούνται εκπομπέ από τα κράτη μελημένα. Ισχύει πολύ έλλειψη διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο ε, τα, εσόδα, τα έσοδα από τι δημοπρασίε χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Και για να πάμε σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να έχουν πιο σαφεί κατευθυντήριε γραμμέ έτσι ώστε τα έσοδα αυτά να χρησιμοποιούνται για δράσει υπέρ του περιβάλλοντο και για να δημιουργηθούν βιώσιμε θέσει εργασία. Για τον κατάλογο τη διαρροή άνθρακα και τα σημεία αναφορά χρειαζόμαστε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση. Το σύστημα που έχουμε το τώρα δεν βασίζεται αρκετά σε συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι δίτο και αυτό που χρειαζόμαστε είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που δεν θα, που δεν θα χρειάζονται τα στοιχεία αναφοράς τα οποία είναι benchmark που προκύπτουν από το 2008 και από την παραγωγή εκεί. Γιατί στις 17 Μαρτίου που είμαστε σήμερα, εγώ είμαι πρώτη γενιάς ε, μετανάστρια από την Ιρλανδία, οπότε σας εύχομαι να ε, τον ε, Άγιο Πατρίκιο σήμερα. Επόμενος ομιλητής. Κύριο Σαπχάουζερ. Πρώτο σχόλιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσατε τους συναδέλφους μου των διαφόρων πολιτικών ομάδων, τις επικρίσεις τους και νομίζω ότι θα τις λάβετε υπόψη. Θα συνεχίσετε τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό είναι σταθερά είτε είστε αποτελεσματικοί και είναι όλεθρο το αποτέλεσμα, είτε είστε αναποτελεσματικοί που είναι επίση όλεθρο το αποτέλεσμα. Θα ήθελα απλώ να πω ότι αν θέλατε λίγο να είστε συνεπεί, θα έπρεπε να λάβετε υπόψη τα σχόλια που έκανε ο συνάδελφο Μαχτά για την προσαρμογή του διοξείδου του άνθρακα στα σύνορα. Αυτό είναι απόλυτη ανάγκη. Δεύτερο σχόλιο. Αν θέλατε να είστε αποτελεσματικοί, δεν θα πρέπει να ασχοληθείτε με τις ε, βιομηχανίες που τις ε, οδηγείται σε μετακατάσταση, ε, άρα περισσότερη ύπανση, αλλά να πάτε και στις θαλάσσιες μεταφορές που ευθύνονται για το 5% των αερίων του θερμοκηπίου. Με την πολιτική σας δεν υποχρεώνεται απλώς τον κόσμο να φύγει και να πάει εκεί που θα ρηπαίνει περισσότερο, αλλά εξαιρείται και τις μεταφορές. Το πρόβλημα για την Ευρώπη, και σας το λέω και είμαι ακράδαντα πεπισμένος και δεν μπορείτε εσείς να αλλάξετε τίποτα σε αυτό, ούτε φταίτε, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η Ευρώπη με δημοκρατικό τρόπο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είπα και στο συνάδελφό σα για το Τίτι που ήρθε να μας μιλήσει. Ο στρατηγός Ντεγκόλ έβλεπε μια Ευρώπη χωρίς κομισιόν και πολλοί από εμά το χαζόμαστε και φανταζόμαστε μια Ευρώπη χωρί την Κομισιόν. Γιατί εσεί καταστρέφετε την Ευρώπη. Εσεί ο ίδιο προσωπικά δεν φταίτε. Σα έχουν βάλει στι ράγε και προχωράτε. Αλλά Κανονικά ήταν ένα μεγαλειώδες, ένα καταπληκτικό εγχείρημα η Ευρώπη και ε, έχει γίνει καταστροφική και σε αυτή την Ευρώπη είμαστε εδώ εμείς για την υπηρετούμε. Ευχαριστώ κύριο Νταν Νίκα. Ευχαριστώ. Καθόμαστε εδώ και συζητάμε για αυτά τα θέματα για από χτες. το απόγευμα έμαθα ότι οι μεγάλες προσδοκίες της Χαλιβουργίας δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Απλώς παρατείνουμε τη διαδικασία αντι-dumping. Δηλαδή όλα αυτά τα περίφημα και τα μεγαλεπίβολα που περιμέναμε δεν έχουν επαλήθευτεί. Το απόγευμα θα γυρίσω στην εκλογική μου περιφέρεια που έχουμε από τα μεγαλύτερα χιτήρια στην Ευρώπη και ε, θα τους πω ότι δεν κάναμε τίποτα, μια τρύπα στο νερό. Ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι το ETS. Σου λέει θα αυξηθεί το τιμολόγιο με μένα ή όχι ε, του ηλεκτρικού. Αυτό τους ενδιαφέρει. Ακούμε διάφορες Παρεμβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενημέρωση, δεν μας λέτε ποτέ αν θα αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Θα γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Αυτό νοιάζει τον κόσμο. Δεύτερον, οι συνάδελφοί μου στη Ρουμανία έμαθαν ότι υπάρχουν τώρα δείκτες benchmarks που δεν ακολουθεί καμία χαλιβουργία και κανένα χιτήριο. Όσο σύγχρονο και να είναι ε, το εργοστάσιο, ε, αυτά τα κριτήρια ποιος τα αποφασίζει για τη βαθμολόγηση. Πρέπει να είναι κάπως ε, ρεαλιστικά αυτά που προτείνεται και όχι τελείως άσχετα με την πραγματικότητα. Έχω συναδέλφους στη Χαλιβουργία που μου είπανε ότι έμαθαν το εξής. Αυτά που εσείς προτείνετε τιμωρούν εκείνους που παράγουν μέχρι τώρα περισσότερο. Παρόλο που το σχέδιο Juncker προβλέπει επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης. Τι θα γίνει τώρα, όταν έχει εργοστάσια που παράγουν στο μέλλον αυτοί θα τιμωρούνται και θα ε, τους επιπλήττουμε. Εγώ τώρα δεν μπορώ να δεσμευτώ για το, ούτε να πω τίποτα για τα ταμεία καινοτομία και εξυγχρονισμού. Έχω συναδέλφου και πάλι από τη Χαλιβουργία που μου λέγουν ότι ποιο εξυγχρονισμό. Αν ε, γίνουν τέτοια πράγματα, εμεί θα καταστραφούμε, θα χαθούμε, θα αφανιστούμε. Τι να εξυγχρονίσουμε. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Βέμπε. Ε, Βέρνε, συγγνώμη. Έχω δύο ερωτήσεις. 50 τομείς λέτε, ενώ σήμερα είναι 75 για το carbon ε, ε, leakage. 175 ήταν στο παρελθόν και τώρα θα γίνουν 50. Πολύ μεγάλη πρόοδος. Ωραία. Είναι πολύ θεωρητικά όμω αυτά που ακούμε. Αυτό που χρειαζόμαστε ω Επιτροπή Βιομηχανία είναι μια δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποιοι θα είναι αυτοί οι 50 κλάδοι, για να ξέρουμε τι γίνεται και να μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση αν είναι θετικό ή αρνητικό για τη βιομηχανία, γιατί είμαστε Επιτροπή βιομηχανία. Να ξεφύγουμε λίγο από το αφηρημένο επίπεδο παρακαλώ και να μπούμε στην πράξη. Κάτι που έχει προβλήματα για μένα είναι τι κάνουν τα κράτη-μέλη με το έμεσο κόστος, γιατί δεν έχουν ενιαία αντιμετώπιση. Ορισμένα κράτη-μέλη το αποζημιώνουν, άλλα πάλι όχι. Χρησιμοποιούν τα έσοδα από το ETS για εξυγίανση του προπολογισμού νομίζω θα πρέπει να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή γραμμή και προσέγγιση. Τα έσοδα από την πώληση των αδειών ETS θα πρέπει τουλάχιστον εν μέρη να ε, χρησιμοποιούνται για την αποζημίωση των εμέσων ε, ε, δαπανών και να γίνεται αυτό με τρόπο ενιαίο κάπως. Θέλω να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ρόιλ. Ευχαριστώ. Άκουσα και εγώ με προσοχή και είπαν όλοι ότι θέλουν να προστατεύσουν το κλίμα αλλά και να μην απειλήσουν πάρα πολύ τη βιομηχανία. Ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε από τον συνάδελφο για τη Ρουμανία, ε, για τη Χαλιβουργία και από την κυρία Βέρνε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε άσκοπα τη βιομηχανία, αλλά αυτά που λέμε είναι λόγια του αέρα. Εάν υλοποιηθεί αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι επιπλέον επιβάρυνση για την Ευρωπαϊκή ε, ε, Βιομηχανία. Τελεία και παύλα και παράγραφος. Αυτό θα αφορά και τη χαλιβουργία ε, και τα τσιμέντα και τα υπόλοιπα. Και όλη μέρα λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερα έσοδα του κράτους για να αντιμετωπίσουμε ε, την κατάσταση και το προσφυγικό. Ε, ας είμαστε ειλικρινείς, να μην λέμε τέτοια πράγματα. Τα κράτη-μέλη, λέει, θέλουν να έχουν υψηλούς στόχους για το κλίμα χωρίς να επιβαρύνει τη βιομηχανία και ο μόνος συνεπής τρόπος είναι ο επιμερισμός των δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποια δικαιώματα που είναι δωρεάν και κάποια άλλα που είναι με δημοπρασία. Τα κράτη-μέλη ε, χρησιμοποιούν, έχει δίκιο κυρία Βέρνερ, τα έσοδα για έχει τρόπους και, και σκοπούς, για να βουλώνουν τρύπες στον προϋπολογισμό. Να τα δώσουν στη βιομηχανία, χρειάζεται βοήθεια. Γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί αντιτίθεται το Συμβούλιο. Γιατί πολλά κράτη-μέλη θέλουν να τα βάλουν στον κορβανά. Ωραίο επιχείρημα. Νόμιζα ότι ήταν κλιματική πολιτική και βιομηχανική και όχι η ταμιακή των κρατών μελών, των Υπουργών Οικονομικών. Αν είχαμε εμεί εδώ το θάρρο να πούμε ότι το 43% και το 57% το μετατοπίζουμε υπέρ της βιομηχανίας, τότε θα κερδίζαμε και πολύ κόπο και πολύ ενέργεια και πολύ χρόνο με τους μικροκαπτάδες για να δούμε ποιο κλάδο της βιομηχανίας μπορούμε να ενισχύσουμε γιατί εδώ πραγματικά διαπληκτιζόμαστε χωρίς ε, κανένα αποτέλεσμα. Να τα πάρουμε από τα κράτη-μέλη, θα τους ε, χάσουν αυτά λίγα έσοδα, δεν πειράζει, αλλά θα βοηθηθεί η βιομηχανία και το κλίμα τελικά. Για να δούμε, το έχουμε αυτό το θάρρος να τα κάνουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Γκερμπράντι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να αναφερθώ στην Φωνή των Παρισίων. Μην υποτιμούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση. Ότι θα κινηθεί ο κόσμος προς μια οικονομία χαμηλή σε άνθρακα. Άρα εκπομπή χαμηλότερων ποσοτήτων άνθρακα στο μέλλον θα κάνει τη βιομηχανία μας πιο ανταγωνιστική. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό και να το εξετάσουμε. μου σημασία είναι να ακολουθήσουν οι επενδύσεις στη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Καρίνς πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την επενδυτική, τη διαρροή επενδύσεων που αποκάλεσε, πώς την αποκάλεσε. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πολιτική για τον άνθρακα σε ποιο βαθμό παίζει ρόλο στη διαρροή των επενδύσεων. Αν δω τις εκθέσεις του ΩΣΑ αναφέρουν ότι εν γέννη στην νομοθεσία περιβάλλοντος ε, επηρεάζεται από την νομοθεσία η ανταγωνιστικότητα και εκεί συμπεριλαμβάνεται και η πολιτική του άνθρακα. Πώς τα βλέπετε εσείς, ερώτηση. Δεύτερο, για τις επενδύσεις. Εξυγχρονισμό, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, το Ταμείο Επενδύσεων. Μπορούμε να επενδύσουμε κάθε ευρώ άπαξ. Άρα χρειάζεται σωστή προσέγγιση. Υποστηρίζω τα όσα είπε το ECR. Πρέπει να θεσπίσουμε αυστηρά κριτήρια για τα ταμεία. Για το Ταμείο Εξυγχρονισμού υπάρχει μεγάλη έλλειψη διαφάνειας. Με τα βίας γνωρίζουμε αν οι επενδύσεις κατά το παρελθόν του Ταμείου Επενδύσεων πήγαν σε τεχνολογία χαμηλού άνθρακα και αν ανταυτού πήγαν σε τεχνολογία υψηλών εκπομπών άνθρακος. Ε, ο κ. Ντελμπέκε ίσως θα μπορούσε να το εξηγήσει αυτό. Αν θα πρέπει να αναμένουμε αυστηρότερα κριτήρια και μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την χρήση των πόρων του Ταμείου Καινοτομίας αλλά επίσης και του Ταμείου Εξυγχρονισμού. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Μπένστεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η διαρροή του άνθρακα είναι σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Χρειαζόμαστε και τη βαριά βιομηχανία στην Ευρώπη στο μέλλον. Συμφωνώ με τον, ε, τον κ. Βλέπουμε κάποιες επιχειρήσεις ε, που έχουν δωρεάν ε, ποσοστώσεις και δεν χρησιμοποιούν και πολλούν τις άδειές τους. Ε, κατά την άποψή μου θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιηθεί αυτό ε, για το Ταμείο Καινοτομιών ή κάπου αλλού. Κατά την άποψή μου ε, είναι θέμα άμεσης κατοικών, κατοικής ενίσχυσης για τις εταιρείε. Κάποιες ε, κάποιες εταιρείες χρειάζονται αυτή την ελεύθερη κατανομή των ε, ποσοστώσεων και δεν λαμβάνουν, άλλες έχουν και δεν τη χρησιμοποιούν. Πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Άλλο που ζητά το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, δεν βλέπω να ζητά άλλο το λόγο. Ίσως να πω εγώ εν συντομία δύο πράγματα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για κάποιες χώρες και για τους πολίτες μας είναι μεγαλύτερη υποστήριξη για τη θέρμανση ε, περιοχών, ε, γενική κεντρική θέρμανση αν θέλετε, ε, αντί να είναι απομονωμένες, μονομενές μονάδες θέρμανσης στα διαμερίσματα, υπάρχει κεντρική θέρμανση, θέρμανση γειτονιών, περιοχών κλπ. Το φυσικό αέριο είναι καλύτερο, φαγματος χάρη από ότι ο άνθρακας για την κεντρική θέρμανση. Αυτό αν εξετάστηκε. Δεύτερον, ελεύθερη κατανομή λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μονάδων παραγωγής για να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης για τους καταναλωτές, για το Ταμείο Καινοτομίας, ε, ποιος θα είναι ο σκοπός του στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος ETS. Για το Ταμείο Εξυγχρονισμού να λάβουμε υπόψη τα δικαιώματα των δικαιούχων χωρών να μπορούν να αποφασίσουν προς ποιαν κατεύθυνση θα κινηθούν οι πόροι. Διαφορετικό από αυτό που έλεγε ο συνάδελφος Herbert Ρόιλ Δηλαδή ότι θέλουν ε, άλλου είδους υποστήριξη. Εδώ είναι διαφορετικό θέμα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν πού θα πηγαίνουν οι πόροι του Ταμείου Εξυγχρονισμού. Στην προσέγγιση μας λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι όσον αφορά τους πόρους και όσον αφορά την τεχνολογία. Αναφέρθηκε αυτό και στη Συμφωνία των Παρισίων προσφάτως. Κύριε Γενική Διευθυντά, μπορείτε να δώσετε απαντήσεις, έχετε κάποια σχόλια να μας ε, παρουσιάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω λοιπόν στις πολύ λεπτομερείς ερωτήσεις ε, που άκουσα ε, ξεκινώντας με πέντε συγκεκριμένα θέματα που θέσατε. Καταρχήν, το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φεύγει κάτι καινούριο. Εμεί ακολουθούμε τι οδηγίε που μα έδωσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Εγκρίθηκε ομόφωνα από όλου τον Οκτώβριο του 2014. Και μπορεί να επαναληφθεί και σήμερα και αύριο στην, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλαμε μια δήλωση για την συμφωνία στο Παρίσι. Οι αρχηγοί κρατών αποφάσισαν πως το σύστημα των ελεύθερων των δωρεάν ε, κατανομών δικαιωμάτων θα είναι ε, το κατάλληλο για να καταπολεμήσει την διαρροή άνθρακα. Και γι' αυτό λοιπόν το επιλέξαμε και δεν επιλέξαμε το άλλο σύστημα γιατί θα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα με τον ΠΟΕ και πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να έχουμε μέτρα για συνοριακά από τη στιγμή που συμφωνήσαμε στο Παρίσι πως ολόκληρη η Σύλλος θα μπορουσαμε αλλωστε να εχουμε μετρα για απο κάποια μέτρα για τον άνθρακα. Δεν λέμε πως όλοι έχουμε φτάσει στο ίδιο σημείο. Όχι. Αλλά θα ήταν πάρα πολύ περίεργο η μεγάλη επιτυχία του Παρισιού το ότι δηλαδή ακολουθούν ε, όλη την ίδια προσέγγιση στον κόσμο, να αντιμετωπιστεί από μια δήλωση δική μας που θα έλεγε ότι θα κάνουμε μέτρα ε, συνοριακά, τα border measures δηλαδή. Τώρα, Είχαμε και το κείμενο των γαλλικών αρχών. Ο κανονισμός ε, για τη ρύθμιση των τιμών δεν συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και έχουμε, και έχουμε την παλιά ΚΑΠ ε, που είχε βασιστεί στον καθορισμό, ε, στον καθορισμό τιμών ε, που τελικά δεν λειτουργήσε και με πολύ συνειδητό τρόπο το αφήσαμε στην άκρη. Η αρχή καρτών και κυβέρνηση υπέγραψε μια δήλωση η οποία πολύ σαφής για το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι πρέπει να κάνει ο νομοθέτης. Μπορεί βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αποφασίσουν κάτι διαφορετικό, αλλά οι οδηγίες που λέγαμε ήταν πάρα πολύ σαφείς για τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα και τη διαρροή του άνθρακα, να σας πω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει απολύτως ότι υπάρχει θέμα ανταγωνιστικότητας. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να εγκαταλείψει την Ευρώπη η βιομηχανία. Όχι γιατί η τεχνολογία είναι πολύ καλύτερη, αλλά και για άλλους λόγους. Στο παρελθόν κάναμε πάρα πολλές έρευνες και δεν υπάρχει τίποτα που να τεκμηριώνει πως υπάρχει διαρροή άνθρακα. Ε, μία ανεξάρτητη πηγή του ΩΣΑ το ε, τεκμηριώνει. Εμείς δεν ήμασταν στη μελέτη αυτοί παρόντες, αλλά δεν υποσκάπτει αυτό το γεγονός πως η διαρροή άνθρακα είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά. Και αυτό κάνουμε εδώ με τους δείκτες αναφοράς, με τους ε, benchmark για την βιώσιμη ανάπτυξη αποφασίστηκαν το 2008 και είπαμε θα αποφασίσουμε μέχρι το 2030. Θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε και αυτό είναι το λάχιστο όσο μπορούμε να κάνουμε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει τεχνολογική πρόοδος η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί γιατί ποια θα είναι η ανταμοιβή σε, σε επίπεδο συντελεστή διορθωτικό ε, διακλαδικό θα βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Γιατί ακόμα και αν το 43% των ε, δικαιωμάτων ε, δοθεί σύμφωνα με αυτό, είναι ένας περιορισμένος, οπότε αν δώσουμε περισσότερα σε κάποιον, τότε αφαιρούνται από κάποιον άλλο. Αυτό υπονοείται. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσους ε, ζήτησαν να τονίσουμε περισσότερο την καινοτομία και το σχετικό ταμείο, γιατί η Ασία αυτή τη στιγμή έχει και παρουσιάζει τεχνολογίες ε, χαμηλής ε, χρήσης άνθρακα. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η τεχνολογία ε, που υπάρχει εκτός Ευρώπης είναι πολύ ανταγωνιστική και ελπίζω πως η Ευρώπη θα μπορέσει και στο γυαλί και στο χάλιβα και στο χαρτί και στα τσιμέντα να διατηρηθεί στην αιχμή του δώρατος της τεχνολογίας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούσαμε και μία ερώτηση για το κατά πόσο η πρόταση για την κατανομή προσπάθειας μπορεί, αυτό νομίζω είναι η ερώτηση της κυρίας Ντελάγκε, για να απαντήσω όχι. Γιατί η αρχηγοί κρατών ήταν πολύ σαφείς. Πώς, θα, πώς θα πρέπει να κατανείμουμε τις προσπάθειες που θα κάνουμε και την ευθύνη που έχουμε ανάμεσα στα δύο συστήματα, δηλαδή το ETS και το effort sharing, οπότε το περιθώριο που υπάρχει και η διαφορά που υπάρχει και δημιουργείται από τα δύο συστήματα δεν είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη στη στιγμή που προετοιμάσουμε την πρότασή μας τώρα για τα έμεσα κόστη. Εμείς προτείνουμε κάποιες διατάξεις σχετικέ με τις κρατικές επιδοτήσεις, κρατικές ενισχύσεις. Έχουμε το έμεσο κόστος όπου η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική στα διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή, άλλο είναι εντατική σε κατανάλωση ενέργειας ε, παραγωγή ε, σε κράτος που χρησιμοποιεί ΑΠΕ ή πυρηνικά και σε άλλο που χρησιμοποιεί ε, ορυκτά καύσιμα, άνθρακα κτλ. Οπότε νομίζω για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το δρόμο των κρατικών ενισχύσεων αναγνωρίζοντας πως είναι περιορισμένες οι ελεύθερες κατανομές και βεβαίως θα πρέπει να ε, προσέξουμε πάρα πολύ στο πώς θα κατανεμηθούν αυτά τα δικαιώματα γιατί ε, αν ανοίξουμε την πόρτα για το κόστος ε, τότε επειδή το κόστος παραγωγής είναι τόσο διαφορετικό ε, για τις εκπομπές στην Ευρώπη που δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Πάντως ελπίζουμε πως οι κρατικές ενισχύσεις θα μας βοηθήσουν στο να τα πετύχουμε. Διαφάνεια, περισσότερη διαφάνεια. Βεβαίως, ενθέρομαι θα το στηρίξω. Έχουμε το Ταμείο ε, Εξυγχρονισμού με το 10C. Περισσότερη διαφάνεια είναι καλή για όλους, είναι καλή για την ανταγωνιστική θέση των οικονομιών μας, αλλά επίσης η διαφάνεια όταν προέρχεται από τα έσοδα, από τις δημοπρασίες, θα πρέπει ε, να ληφθεί δεόντως υπόψη. Οι δημοπρασίες αυτές είναι σημαντικές. 60-70 δις υπολογίσαμε τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο, οπότε πολλά λεφτά. Και πού θα πάνε. Πώς θα χρησιμοποιηθούν. Ίσως για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τα μέτρα εκεί. Είτε για την παρότρινση χρήσης ενέργειας ε, χαμηλής ε, κατανάλωσης άνθρακα. Θα μπορούσαν δηλαδή να κάνουν πολλά τα κράτη-μέλη. Μπορεί να πάνε στην τεχνολογία ΑΠΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία. Αλλά η περισσότερη διαφάνεια σίγουρα θα μας βοηθήσει ως πρώτο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και για την τηλεθέρμανση να σας πω πως ο εξυγχρονισμός, το Ταμείο Εξυγχρονισμού είναι η ιδανική πηγή και να έχουμε τέτοιου είδους ε, επενδύσεις. Αλλά και τα έσοδα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούν για την τηλεθέρμανση. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα αυτό. Όσοι έχουν τηλεθέρμανση ξέρουν πως έχουν ένα πολύ ε, καλό εργαλείο ε, στα χέρια τους. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή βασίζεται υπερβολικά στα ορυκτά καύσιμα, αλλά με μια μικρή αλλαγή θα μπορούσε να φέρει μεγάλα πλεονεκτήματα γενικότερα σε προσπάθεια που κάνουμε ε, στη μείωση των εκπομπών ανακράτως μέλος. Ευχαριστώ πολύ και, και διευθυντά σαφέστατες οι απαντήσεις σας. Αν παρελήφθη απάντηση, δεν ξέρω. Σύντομα, κύριε Γενική Διευθυντά, λέει ο Νίκα, μία ερώτηση. Ο τη της μεταρρύθμισης θητείας στην τιμή τη ενέργειας, Ποιο θα είναι. Να περιμένουμε αύξηση και αν ναι, πόσο. Μείωση, αν ναι, κατά πόσο. Καλώ 10 δευτερόλεπτα ερώτηση-απάντηση. Σας παραπέμψω στην αξιολόγηση αντικτύπου όλα εξαρτώνται με το πώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. Αν παράγεται υδροηλεκτρικά με πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, έχουμε μηδενική επιρροή στην τιμή. Αν έχουμε ορυκτά καύσιμα, έχουμε αποτελέσματα στην τιμή μεγαλύτερα. Αυτό είναι και ο σκοπό. Να δώσουμε κοίτα επιχειρήσει να μειώσουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Μία ερώτηση ο καθένα. Δεν θέλω να επιμένω, κύριε Γενική Διευθυντά οι τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξη Ανοικοδόμηση αρνούνται επενδύσεις, προσπαθούν να δώσουν κίνητα στα κράτη-μέλη να αλλάξουν την παραγωγή ενέργειας από ρηχτά καύσιμα σε μη ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας. Άλλη ερώτηση, πρέπει όλοι να μπορείτε να μιλήσετε. Έχετε πολλά λεπτά μπροστά σα, ε, Φρέντερικ, δεν είναι για Έχετε χρησιμοποιήσει πολλά, ο κ. Μαρτέν. Κύριε Διευθυντά, Όταν λες ένα ψέμα και το αναλαμβάνει, δεν γίνεται αλήθεια αυτό. Γιατί είναι κατά του ΠΟΕ η προσαρμογή στα σύνορα. Θα πρέπει να είναι όλοι ε, στην ίδια μοίρα. Δηλαδή ο ΠΟΕ τι ε, προωθεί την ανισότητα. Ναι. Τέλος του γύρου των ερωτήσεων των 10 δευτερολέπτων. Το λόγο έχει ο εισηγητής μας, ο κύριος Φέντερλε. Στο τέλος προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Κοιτάξτε, όλοι οι σκιώδεις με το ίδιο θέμα και τον ίδιο στόχο. Ποιος είναι? Εκείνοι που είναι στο 10% που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις να έχουν τις δωρεάν άδειε. Αυτό που συνέβη είναι ότι την αρχή ο διορθωτικό ε, συντελεστής ε, λειτουργήσε και επέφερε αλλαγές στην αγορά, στους υπολογισμούς και στις δωρεάν ε, χορηγήσεις αδειών. Το βασικό θέμα είναι να έχουμε την κατάλληλη προσέγγιση. Αυτός είναι ο σκοπός της Επιτροπής Ήτρε. Στο Παρίσι. Περίμενε έστερα για απάντηση. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδράζεται, το ETS εδράζεται, επί των στόχων για το κλίμα που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν χρειάζονται μεγάλες προσαρμογές στην πρόταση μετά τη Συμφωνία των Παρισίων. Συμφωνώ με αυτή τη βασική άποψη. Δεν έχουμε νέους υπολογισμούς, έχουμε νέες προτάσεις. Αυτές θα είναι η βάση των εργασιών μας. Και για το μέλλον. Τούτου λεχθέντος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αργότερα ίσως πρέπει να γίνουν προσαρμογές και ίσως θα πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση να συμμορφωθούμε με την COP21. Τώρα, σε αυτή τη φάση, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να υπολογισμοί. Συνεχίζουμε με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουμε από αυτή της βάσης της εργασίας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε, για τα σχόλιά σας. Θέλετε να απαντήσετε ίσως στο τελευταίο θέμα. Πολύ γρήγορα. Δεν νομίζω ότι ο ΠΟΕ τοποθετείται επί ισότητας, έχει σαφείς κανόνες και προσανατολισμούς για τη διοργάνωση του παγκοσμίου εμπορίου. Σέβεται τις πολυμερείς συμφωνίες. Στο Παρίσι απλώς συμφωνήσαμε, όλος ο κόσμος συμφώνησε. Προσπαθώ να σα εξηγήσω ότι ήταν πολύ παράδοξο να πούμε ζήτω συμφωνεί όλος ο κόσμος στην αρχή και τώρα να αρχίσουμε νέα διαδικασία στον ΠΟΕ για περιορισμό του εμπορίου. Οι ίδιοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μας είπαν αν υπάρχουν συνέπειες για το εμπόριο χρησιμοποιήστε τις δωρεάν άδειες γι' αυτό. Ε, συνάδελφοι, ήταν πολύ σημαντική συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι και στο μέλλον θα έχουν έτσι τα πράγματα και θα διεξαχθούν συζητήσεις στην Επιτροπή μας. Καλό προσωπικά τον συνάδελφό μας, τον Ντάνκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι ο βασικός υπεύθυνος να έρθει για να ακούσει τις απόψεις μας. Θα πρέπει να βρούμε συμβαστική λύση επί πολλών θεμάτων οι δύο επιτροπές. Ευχαριστώ όλους σας. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, σας ευχαριστώ πολύ για την πληρέστατη παρουσίαση του θέματος και την προσέγγιση σας και συγχαρητήρια για το έξοχο έργο που επιτελείτε. Okay. Uh, Renewable Energy Progress Report. Uh, Επόμενο σημείο. Παλώμα Λόπεθ Βερμέρο, συγκεκριά, της Γκουε. Στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια επισκόπηση της οδηγίας, ανα, ε, της οδηγίας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το τέλος του έτους και ποιους στόχους έχουμε θέσει μέχρι τέλος ε, του 2020 τουλάχιστον 20% και 27 περίπου μέχρι το 2030 άρα είναι πολύ σημαντική η έκθεση από αυτή την πλευρά η συγγήτρια, ε, κυρία Λόπες Μπερμένο, να μιλήσει για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους τους παρόντες για τη δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε πριν τη συνεδρίαση με τους σκιώδεις συγητές για να ανταλλάξουμε απόψεις για την έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία ε, για την ταχύτητά της έτσι ώστε να έρθει γρήγορα ένα προσχέδιο έκθεσης και μάλιστα στα χέρια των εισηγητών των σχεδόν κάθε πολιτικής ομάδας. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να στείλει το Κοινοβούλιο μας ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ΑΠΕ με ορίζοντα το 2030 η Επιτροπή μας που είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας θα πρέπει να ε, συνεργαστεί χέρι-χέρι με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Από τη μία τι διακυβεύεται, η δυνατότητα της Ευρώπης να εξακολουθεί να είναι ηγετική στην ε, εξέλιξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να διατηρήσει ε, το πλεονέκτημα αυτό που έχει, ε, το βιομηχανικό και να εξασφαλίσει και την ενέργεια. Γενικότερα υπάρχει όμως και μια παγκόσμια πρόκληση που είναι να προσαρμοστούν οι οικονομίες μας στις πιο απαιτητικές προδιαγραφές για το περιβάλλον έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την κλιματική ε, αλλαγή και να εξασφαλίσουμε το μέλλον των επερχομένων γενναίων. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω ε, σε θεμέλια που ήδη υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να εφευρίσκουμε τον τροχό κάθε φορά. Ε, στόχοι δεσμευτικοί, εθνικά σχέδια και μηχανισμοί ελέγχου έχουν οριστεί και ήταν και αποφασιστική σημασία έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να τηρήσει το 2020 το στόχο του 20%. Θυμίζω ότι ο στόχος αυτός αφορά την κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει και τις υποστήριξη του Κοινοβουλίου στο παρελθόν. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και τους στόχους αυτούς για το μέλλον. Σήμερα είναι πολλά εκείνα τα κράτη-μέλη που καλύπτουν τους εθνικούς στόχους ήδη με τις προσπάθειές τους. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η σταθερότητα των μηχανισμών στήριξης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρειάζεται ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέτρα εκείνα που τιμωρούν την ίδια κατανάλωση ή ε, την αναδρομική ε, στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως σημαίνει στην Ισπανία, είναι παραδείγματα ε, κακής ε, πρακτικής και θα πρέπει να αποφεύγονται αν θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη του κλάδου. Και γι' αυτό το λόγο και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Άλλωστε η ομάδα μας ε, θα δώσει προσοχή και στα κοινωνικά θέματα με τον εξή διπλό τρόπο. Θα πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση σε ένα ενεργειακό μοντέλο που θα βασίζεται στη ΣΑΠΕ με στόχο ε, μεταξύ άλλων να καταπολεμήσει την ενεργειακή ένδυα και να υπάρχει ένας εκδημοκρατισμός στην ενέργεια. Δηλαδή τα νέα συστήματα ε, ρύθμισης ή παραγωγής δεν θα πρέπει να αυξάνουν το κόστος για τις ε, οικογένειες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Εμείς πιστεύουμε ότι τα λογικά συστήματα παραγωγής και ενεργειακής απόδοσης θα είναι κρίσιμα στο μέλλον, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ανεξαρτησία για συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στο ίδιο το ενεργειακό τους μοντέλο. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Το δεύτερο είναι το εξής. Γίνονται διαστατικές αλλαγές με τις ΑΠΕ και αυτό απαιτεί προφανώς ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων όταν καθορίζονται τα εθνικά ενεργειακά σχέδια και όταν πρέπει να προσαρμόζεται το εργατικό δυναμικό. Εμείς θέλουμε να δημιουργούνται ποιοτικέ θέσει εργασία στον κλάδο αυτό. Το κείμενο είναι σύντομο, είναι διαρθρωμένο και δομημένο με απλό τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν περισσότερες από τις ιδέες των άλλων πολιτικών ομάδων. Δυστυχώς πιέζει ο χρόνος, αλλά είμαι πεπισμένη ότι αυτό δεν θα αποτελέσει και μεγάλο εμπόδιο για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά για συμβαστικές τροπολογίες. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφος Μπένστεν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Λόπεθ και τους σκιώδης ηγητές συναδέλφους μου για την ανταλλαγή απόψεων που ήταν σύντομη, αλλά έλαβε χώρα από το θέματος. Θα ήθελα να τονίσω κάποια βασικά απορίσματα της ανακοινώσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που νομίζω ότι πρέπει να σημειωθούν στην έκθεση πρωτοβουλίας μας. προσπαθούμε να πετύχουμε το στόχο του 20%. 5 από 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως αναμένεται να πληρούν τα κριτήρια του 2020. 19 από τις 25 χώρες αυτές αναμένεται να ξεπεράσουν τους στόχους. Ο στόχος των μεταφορών έχει μείνει πίσω. Ο μέσο όρος της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι 5,7%. Ήδη επέσα στην προσοχή της εισηγήτριας κάποιες βασικές στοιχές για τους σκοπούς της εκθέσεως για το σκοπό της σημερινής συζητήσεως θα ήθελα να θέσω κάποιες βασικές πτυχές και το ΕΛΚ βεβαίως υποστηρίζει τι πηγές πηγέ ενεργεία. Αναγνωρίζουμε ότι είναι ο αποτελεσματικότερο τρόπο για να μειώσουμε την εξάρτηση από τα ρηχτά καύσιμα, ένα από τους τρόπους, και να μειώσουμε την εξάρτηση από εισαγωγές και να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές ανθρακώ. Αναγνωρίζουμε ότι τις πηγές πηγέ τη ενεργεία ενώσιμες πηγές ενέργειας τονώνουν τη βιωσιμότητα, εξαγωγέ, ανάπτυξη, απασχόληση, έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά με αυτό τονίζουμε ότι θα πρέπει η έκθεση να αντικατοπτρίζει τη σημασία τη ποικιλομορφία όσον αφορά την ενέργεια. Για το ΕΛ και είναι εξίσου σημαντικό η έκθεση σαφώ να δηλώνει ότι οι εθνικέ αρμοδιότητε για το ενεργειακό μείγμα πρέπει να διαφυλαχτούν. Συντάσσοντας την έκθεση θα πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε και τι κεντρικέ προτεραιότητε για τι ανανεώσιμε πηγές ενέργεια όπως καλύτερη επικαιροποίηση της αγοράς ούτε ώστε να λαμβάνει υπόψη τη χρήση ανασύμων πηγών ενέργειας. Είναι σημαντικό για τις ενεργειακές τιμές στην ε, ε, Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητα αυτής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους και την ανταγωνιστικότητα των ανεσίμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμες προπτικές για τις επενδύσεις. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για τη μετώπιση ε, της του τομέα των μεταφορών και που χρειάζεται πραγματικά πρόοδος του, του λεχθέντος. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε το να κατηγορούμε κάποιες χώρες καθώς προχωρούμε προς τους στόχους του 2020. Ε, γενικά προχωρούμε προς τους στόχους. Θα πρέπει η έκθεση να παραμείνει εντός θέματος. Επαναβάνονται κλασικά ζητήματα που είναι επίμαχα ε, και που εξυπηρετούν εθνικά συμφέροντα. Όμως είναι και σήμος σημασίας για την επιτυχία της εκθέσεως να έχουμε συγκεκριμένο στόχο ε, της εκθέσεως, δηλαδή είναι επίτευξη στόχο 2020 συστήνουν να μην προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει αναθεώρηση τι οδηγίε ενώσιμε πηγέ ε, ενέργεια εν ώψη των συζητήσεων του φθινοπόρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπένσον. Εκ μέρου των σοσιαλιστών, Σάμπα Μόλναρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Συγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι. Κατά την άποψή μου, το θέμα των ανεωσίμων δεν αφορά κάτι ιδεολογικό ή πολιτικό αλλά κοινωνικο-οικονομικές πτυχές. Οι ενώσιμες πηγές ενέργειας δεν καταλήγουν μόνο σε καθαρό περιβάλλον, δεν είναι μόνο θέμα πρασινίσματος, μπορεί να προσμετρηθεί επίσης σε εκατομμύρια νέων ποιοτικών θέσεων και τεχνολογική καινοτομία και ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη. Και γι' αυτό αυτή η έκθεση είναι σημαντικότατη. Συνάδελφοι, έχω κάποιες προτάσεις σχετικά με το σχέδιο εκθέσεως, διότι είμαι σκιώδης συγητής και υπόσχομαι ότι θα είμαι σύντομος. Καταρχάς, όπως αναφέρεται στην έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεσμευτική στόχη ήταν βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη δυνατοτήτων χρήσεων ανανεσίμων πηγών ενέργειας στα κάτι μέλη και, στο, και δημιούργηκε βεβαιότητα για τους επενδυτές λόγω των στόχων και αυτό θα ενθαρρύνει και περαιτέρω επενδύσεις ανανεώσιμε στο μέλλον. Έτσι περαιτέρω αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και στόχοι μη δεσμευτικοί τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως που τέθησαν το 2009 αλλά εκεί δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος. Ήταν ο τομέας της ενεργειακής απόδοσης αντιθέτω δεσμευτικοί στόχη στον τομέα των ανανεωσίμων επέφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα. Πιστεύω συνεπώ θα πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει εθνικού δεσμευτικού στόχου και μετά το 2020 και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό των ανοσίμων από το 27% μέχρι το 2030. Δεύτερον, στην έκθεση θα πρέπει να εστιαστούμε επί διαφόρων εμποδίων που εμποδίζουν τον επιμερισμό, την αύξηση των ε, χρήσεων ανενοσύμων πηγών στα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα διοικητικά εμπόδια και κάποια τέλη που είναι επιβλαβή για τις ανανεώσιμες και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τα δίκτυα διότι σε πολλά κράτη-μέλη βλέπουμε ότι δεν μπορούν να δεχτούν ε, ισχύ που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Χρειάζεται ε, εξυγχρονισμός των δικτύων των ενεργειακών και αυτό θα πρέπει να τονιστεί. Πρέπει να τονίσουμε και την ενεργειακή, την αποθήκευση ενέργεια, εφή μέτρηση της ροής ενέργειας κλπ. Θέλουμε σύγχρονες λύσεις σε μια σύγχρονη εποχή. Μιλώντας για εμπόδια θα πρέπει να τονίσουμε ότι η τρίτη γενιά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Ε, η κεντρική παραγωγή ενέργειας, αυτοπαραγωγή είναι κάτι που θα κάνει πιο φθηνή την ε, τιμολόγηση, πιο φθηνό το κόστος της ενέργειας στα νοικοκυριά. Ευχαριστώ λοιπόν ε, του Σκιώδης ε, για τη βοήθεια, για, για τις συζητήσεις, για την έκθεση. Στο τέλος πιστεύω ότι θα πετύχουμε μια ισορροπημένη έκθεση που θα τύχει υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ εκ μέρους του ECR η κυρία Έλεν Βαν Μπόλσιλτ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή εισηγήτρια, Μέχρι το τέλος της θητείας θα μας απασχολήσει πολύ στην Επιτροπή μας το θέμα των ΑΠΕ. Με πολύ μεγάλη προσοχή διαβάσα την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο έκθεσης της ηγήτριας που το λάβαμε και συμφωνώ ε, και θα κάνω και προτάσεις. Κρίμα που σήμερα δεν μπορούμε να μπούμε στην ουσία ε, να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης. Θα περιοριστώ στην ε, αντίδρασή μου ε, στην ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως και όδηση συγγήτρια της ομάδας μου θέλω να τονίσω τρεις προτεραιότητες που έχουμε εμείς. Το πρώτο είναι η ενεργειακή απόδοση. Ενδιαφέρουσα τα, η έκθεση που ακούσαμε χτες, η παρουσίαση και τη χθεσινή συζήτηση τη θυμάστε και φαίνεται όλο και περισσότερο ότι για την ενεργειακή απόδοση χρειαζόμαστε ακόμα πολλή δουλειά. Χρειάζεται καλύτερη αντιμετώπιση της ενέργειας που έχουμε και εξοικονόμηση. Ε, στο Βέλγιο ε, που έχουμε περιορισμένες δυνατότητες παραγωγής ΑΠΕ ε, πρέπει να ποντάρουμε στην ενεργειακή απόδοση, στην εξοικονόμηση δηλαδή ενέργειας. Δεύτερον, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι μεν, πλην όμως να αναγνωρίζουμε και τις πραγματικότητες. Εγώ είμαι από τη Φλάνδρα και δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες, είναι περιορισμένη η δυνατότητα παραγωγής ΑΠΕ, δεν έχουμε πολύ ε, ε, χώρο, μεγάλη επιφάνεια, δεν έχουμε πάρα πολύ ήλιο και τέτοια πράγματα. Οπότε ε, πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε ανεμογεννήτριες στη θάλασσα που είναι ακριβή επένδυση και μέχρι το 2030 θα πρέπει να έχουμε πιο αποτελεσματικό ε, τρόπο στη διαχείριση της ενέργειας. Και ένα τρίτο στοιχείο που δεν είναι λιγότερο σημαντικό, ακόμα και αν το λέω τελευταίο, είναι καλύτεροι κανόνες και ρυθμίσεις για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ΑΠΕ χρειάζεται μια ενεργειακή αγορά με καλύτερες διασυνδέσεις και ε, πιο γρήγορη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Δυστυχώς ε, είμαι υποχρεωμένη να διαπιστώσω ότι παραμένουν πάρα πολλοί ε, διοικητικοί και τεχνικοί κανόνες που μας δυσκολεύουν τη ζωή. Με αυτές τις τρεις προτεραιότητες ε, προσβλέπω στη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους υπολείπους και όλους εισηγητές. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλντε. Γκερμπράντι. Συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τα καλά μαντάτα. Χθε στους Financial Times είδατε στις πρώτες σελίδες ότι σύμφωνα με το Διεθνή, Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας είχαμε μείωση της χρήσης του άνθρακα και χρήση των ΑΠΕ αυξανόμενη. Και γι' αυτό είχαμε χαμηλότερες εκπομπές διεξιδιού του άνθρακα στον κόσμο. Αυτά είναι τα καλά μαντάτα. Οι ΑΠΕ παίξαν σημαντικό ρόλο τα κακά μαντάτα. Δυστυχώς στην Ευρώπη βλέπουμε ότι οι επενδύσεις στις ΑΠΕ μειώνονται. Το 2015 μειώθηκαν κατά 18% και αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό και είναι κάπως αντίθετο με έναν από τους δέκα πολιτικούς προσανατολισμούς του Πρόεδρου Γιούκεν. Είπε ότι θέλει η Ευρώπη να γίνει ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη χρήση των ανανεωσίμων. Στην έκθεση αυτή πρέπει να πω ότι η γέννη εικόνα φαίνεται αρκετά καλή. Είμαστε στη σωστή πορεία για τους στόχους του 2020. Ανησυχώ για κάποιες χώρες, το Λουξεμβούργο, η χώρα μου, η Ολλανδία με ανησυχεί και κάποιες άλλες όπως η Γαλλία, το Ναμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Σίγουρα λοιπόν θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες όχι μόνο για να πετύχουμε τους στόχους του 2020 αλλά να επιτύχουμε στο τέλος και μεγαλύτερη πρόοδο. Ήδη αναφέρθηκε από άλλους συναδέλφους ότι υπάρχει, ότι έλλειψη, υπάρχει έλλειψη δεσμευτικών στόχων στο μέλλον. Η έκθεση πρόοδου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι είναι επωφελή η δεσμευτική στόχη και απευθύνει η έκκληση να συνεχίσουν οι δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ. Σημαντικό ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί σταματήσατε. Τέλος, Πρόεδρε. Όταν μιλάμε τη βιομηχανίας παραπονούνται για δύο πράγματα για τις ΑΠΕ. Πρώτα απ' όλα θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη ανανοσίμων πηγών ενέργειας. Δεν χρησιμοποιούν τις ΑΠΕ πλήρως και δεν υπάρχουν ποσότητες επαρκής. Δεύτερον, διαμαρτύρονται για έλλειψη διασυνοριακής συνεργασίας Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ. Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο εδώ και δύο χρόνια θέτησε ένα ψήφισμα που ανέφερε ότι όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνονται επί Ολλανδικού εδάφους για τις ΑΠΕ και όχι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό αντιβαίνει πλήρως όχι μόνο την ευρωπαϊκή ιδέα της Ενεργειακής Ενώσεως αλλά και είναι ανόητος τρόπος να είναι κανείς αποδοτικός αυτό το κόστος. Τέλος, ε, Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι από ό,τι τώρα. Αν δείτε το όλο ιστορικό της μελέτες της Διεθνής Υπηρεσίας Ενέργειας και είναι από τους πιο βασικούς θεσμούς για την ενέργεια. Ιστορικά υποτιμούσαν την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Και όχι μόνο λίγο, αλλά έπεφταν δραματικά έξω. Δεν υπάρχουν αρνητικές πτυχές των ΑΠΕ στο μέλλον είναι πιο καθαρές πηγές, γινόμαστε εξάρτητοι και είναι και πιο φθηνή πηγή ενέργειας στο μέλλον. Ας συνεχίσουμε και ας μάθουμε από τα μαθήματα που περιγράφονται σε αυτή την έκδοση. Ευχαριστώ κύριε Γκερμπράντι. Είχαμε τέσσερις σκιώδεις εισηγητές που μίλησαν για τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες. Ο κ. Μπλάνκο Λόπεθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος να συγχαρώ καταρχήν τον εισηγητή. Είναι πολύ σφροπημένη αυτή η έκθεση και που στιμαχίζει υπέρ του ΑΠΕ. Το, συγγνώμη. Δεν σας είχα δει, με συγχωρείτε, αλλάζω τη σειρά. Λοιπόν, εσύ συνεχίστε. Συχηματίζει λοιπόν υπέρ των ΑΠΕ και επίσης αναφέρεται σε καταστάσεις που θα εγγυηθούν την νομική βεβαιότητα έτσι ώστε να μην έχουμε το θέμα της αναδρομικότητας όπως συνέβη σε κάποιες χώρες όπως η Ισπανία που αμφισβήτησαν με τον τρόπο αυτό κάποιες επενδύσεις και έφεραν μεγάλη αστάθεια. Η έκθεση η οποία προέκυψε από τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως είναι υπεραισιόδοξη και έρχεται σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν σε κάποιες χώρες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία δημιουργούν αστάθεια και αβεβαιότητα για να τα λάβει υπόψη ο συγητής. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως Πολωνία, Ουγγαρία ενδεχομένω δεν θα καταφέρουν να εκπληρώσουν υποχρεώσει. και λέει θα πρέπει η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία θα πρέπει να αξιολογήσουν τι πολιτικέ του. Αυτό χωρί να λάβουν υπόψη τι νέε καταστάσει όπω η ενεργειακή μεταρρύθμιση στην Ισπανία με 0 ε, ΜΒ το 14-15 νέα ΜΒ ή την ε, ε, ε βούληση της πολωνικής κυβέρνησης. Αυτά είναι κρίσιμα σημεία για να εξασφαλίσουμε το κατά πόσο θα ε, καταφέρουμε εμείς τους ε, στόχους του 2020. Ούτε λαμβάνει υπόψη την οικονομική κρίση γιατί ε, έχουν εθιγεί και οι ΑΠΕ, ούτε κοιτάει τα εναλλακτικά σενάρια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα από συζήτηση, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και που θα μας κάνουν λιγότερο αισιόδοξου σίγουρα. Επίσης υπάρχει ένα είδος ε, υπερβολικής ε, αυταρέσκειας ε, και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει πιο ρεαλιστική ανάλυση των δικών της της πράξεων και δεν έχει και τα εργαλεία για να, για να τιμωρεί τους όσους θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους τους οποίους έχουμε όλοι υπογράψει. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ο κύριος Γιαβόρ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ και λυπάμαι που καθυστέρησα γιατί ήμουνα σε συζήτηση στην Επιτροπή ΕΜΒΗ για την ανακοίνωση της ε, Κομισιόν για τα αποτελέσματα της 21 και σχετίζεται πολύ στενά ε, με το δικό μας θέμα. Στην ΕΜΒΗ ήταν σαφές πως οι δικές μας δεσμεύσεις αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκές για να ε, πετύχουμε τους στόχους που έχουμε στη Συμφωνία του Παρισιού και θα πρέπει να τους ξαναδούμε όπως και τις δεσμεύσεις μας και βέβαια να συμπεριλάβουμε και το θέμα με τις ανανέσουμες πηγές ενέργειας για να εκπληρώσουμε τα όσα συμφωνήσαμε στο Παρίσι, πολλά θα πρέπει να κάνουμε με τις ΑΠΕ και η γενικότερη προσπάθεια είναι να έχουμε 100% ΑΠΕ, αυτά ως οικονομική βάση το 2020. Για να συμβεί όμως αυτό έχουμε ακόμα πολλά βήματα. Για να αναφερθώ στα πιο κρίσιμα σημεία, λαμβάνοντας υπόψη και το σχέδιο έκθεσης που έχουμε είναι πολύ ε, θετικό, να κάνουμε όμως κάποιες ε, παρατηρήσεις για να συμπληρωθεί Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ με τον κύριο Γκεμπράντη. Εάν δεν υπάρχουν υποχρεωτικοί στόχοι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Η εμπειρία των τελευταίων ετών μας οδηγούν στο εξή συμπέρασμα. Ακόμα και για την ενεργειακή αποδοτικότητα και για άλλου κλάδου, σχεδόν όλε οι επιτυχίε μας απορρέουν από υποχρεωτικούς στόχους. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτοί οι υποχρεωτικοί στόχοι σε ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο να συνεχίσουν να υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να αυξήσουμε το στόχο μας. Το 27% είναι σε ΑΠΕ, είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο χρειαζόμαστε για το 2030 για να είμαστε πράσινοι, βιώσιμοι. Και ας είμαστε ειλικρινείς. υπολείπεται και της πραγματικότητας στην αγορά. Εάν δεν κάνουμε κάτι πολύ αποτελεσματικό, ο κλάδος να πέσει στην Ευρώπη θα φτάσει, το 23-24% στο 2020 και άλλα 3% για να φτάσουμε το 27% μέχρι αργότερα, αλλά η αγορά έχει ξεπεράσει κατά πολύ στην πραγματικότητα του στόχου μας και θα πρέπει να τους αναβαθμίσουμε. Δεύτερον, τα σχέδια δράση στα εθνικά για τις ΑΠΕ. Είναι αδύναμα. Και θα πρέπει να ελέγξουμε το εξή. Τα κράτη-μέλη όντω σέβονται τι απαιτήσει που έχουν στα εθνικά σχέδια δράση για τι ΑΠΕ. Εφαρμόζονται. Άραγε. Επίσης, μικρές τοπικέ ε, κοινότητες, καταναλωτές, και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση, οι τοπικές κοινότητες και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν ένα ζωτική σημασία ρόλο να παίξουν για να γίνουν πιο πράσινες, πιο βιώσιμες, πιο ανανεώσιμες και οι καταναλωτές ή οι παραγωγοί που ήδη παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθούν, να στηριχθούν έτσι ώστε να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση με ρυθμιστικό τρόπο, κανονιστικό τρόπο αλλά και μέσω επιδότησης τέτοιων, είδων, τέτοιων προσπαθειών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. στρατηγική κατεύθυνση προς τις ανανεώσιμες έχει φέρει μεγάλα πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα στο μεταβλητό κόστος. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα θέσουμε το σωστό πλαίσιο στο μέλλον ε, με τρόπο ανταγωνιστικό. Βέβαια, έχουμε συγκριόμενους στόχους στα υδροελεκτρικά εργοστάσια, για παράδειγμα. Με την οδηγία πλαίσιο για τα είδετα, αφενός, έχουμε πάρα πολύ μεγάλους περιορισμούς στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και από την άλλη τίθεται το ερώτημα πώς θα έχουμε μια αμοιβαία υποφελή κατάσταση. Το άλλο που θέλω να πω είναι η αποθήκευση ε, της ε, υδρο, ε, υδραυλικής ενέργειας μάλλον Ε, ηλιακή και ολική ενέργεια δεν ε, ε, υπάρχουν όποτε θέλουμε. Έχουμε ήλιο το καλοκαίρι και άνεμο τον χειμώνα, αλλά υπάρχουν και περίοδοι χωρίς ηλιοφάνεια και χωρίς άνεμο. Τι θα κάνουμε τότε. Δεν θα πρέπει κάπου στις Άλπεις να έχουμε ταμιευτήρες νερού για να εξοικονομούμε, να αποθηκεύουμε νερό για να το χρησιμοποιούμε σε υδροελεκτρικά εργοστάσια. Έτσι δεν είναι. Αυτό όμως θα σήμαινε ότι και το ανώτατο όριο των τιμών θα πρέπει να ε, αξιολογηθούν γιατί μπορεί να είναι ένα εμπόδιο για επενδύσεις και χρειαζόμαστε ε, ανάλογους δείκτες και ανάλογες κινήσεις και στα χρηματιστήρια. Ευχαριστώ κύριος Μπενίτο Φουλουάδα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, εγώ θα είμαι σύντομος. Η συνάδελφος Λόπεθ, ε, η συγκήτρια, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι και είναι απαραίτητο να αυξηθεί το ποσοστό των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα για να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή. 30% προτείνει το Κοινοβούλιο για το 2030. Θα πρέπει αυτή η πρόταση να διαβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αρχίσει ένας προβληματισμός μήπως χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξους στόχους από τους σημερινούς. Επίσης κάτι που είναι πολύτιμο είναι αυτά που λέει η έκθεση για την ε, αποκεντρωμένη συμμετοχική και δημοκρατική διαχείριση και τις δημόσιες επενδύσεις για να βελτιωθούν οι μέθοδοι παραγωγής και να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια. Είναι στόχος μας και αυτός και ανησυχία που τελευταία ε, είναι όλο και πιο παρούσα και στις συζητήσεις μας εδώ και στην κοινωνία γενικότερα. Ε, ελπίζω η συγγήτρια να λάβει υπόψη αυτά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε να υπάρχουν εμπόδια ούτε διοικητικά ούτε οικονομικά. Δυστυχώς στην Πολωνία και την Ισπανία βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει και παρεμποδίζεται η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Ντοβιντούνης από τη Γενική Διεύθυνση, μάλλον, ο, συγγνώμη, τμήματάρχης από την ε, αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα εκ μας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαριστώ τα μέλη την κυρία Λόπες ε, για το σχέδιο εκθέσεως που παρουσιάστηκε σήμερα και την ευχαριστώ για τις πολύ επικοδομητικές απόψεις. Μάλλον ευχαριστώ όλους που εξέφρασαν θετικές απόψεις στην αίθουσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι περνάμε μια πολύ σημαντική εποχή για την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Απορεί και από την πρώτερη συζήτηση αυτό. Λοιπόν, είναι μια ήσυχη επανάσταση που λαμβάνει η χώρα και διαμορφώνεται. Η Ευρώπη κινείται προς ένα σύστημα ενεργειακό με χαμηλή εκπομπή άνθρακα, ένα ενεργειακό σύστημα που συνεχώς βασίζεται στις ΑΠΕ και η ενεργειακή απόδοση παίζει έναν πολύ κεντρικό ρόλο. Το αναφέρει και το σχέδιο έκθεσης. Όπως σωστά ανέφερε και το μέλος του Ευρωκοινοβουλίου. Η συμφωνία COP21 έδωσε νέα όθηση στο κίνημα και στο Παρίσι αναγνωρίστηκε ο συσχετισμός μεταξύ ενεργειακού τομέα που είναι τα δύο τρίτα τον υπεύθυνο για, τον εκπο, για τις εκπομπές και το στόχο που έχουμε το κλίμα και είναι η ώρα για να αντιμετωπιστεί πραγματικότητα. Βλέπουμε ότι η ΑΠΕ και η ενεργειακή απόδοση πράγματι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις εκπομπές. Βεβαίως δεν έχουν μόνο συνέπειες για το περιβάλλον, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, ανάπτυξη, ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια, μείωση των εισαγωγών. Αυτό είναι το πλαίσιο. Η Ενεργειακή Ένωση θα χρειαστεί μια μεταρρύθμιση του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε αυτό συμπεριλαμβάνει 27% απέ στο ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2030 αυτό είναι 50% τουλάχιστον ΑΠΕ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Και από εθνικούς δεσμευτικούς στόχους κινούμεθα προς δεσμευτικούς στόχους της Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030. δημιουργούνται νέα προβλήματα και νέες ευκαιρίες όμως για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και θα επενδύσουν περισσότερο στις ΑΠΕ. Υπό την προπόθεση τα κράτη-μέλη θα εφαρμόζουν εθνικέ πολιτικέ που προστατεύουν του επενδυτέ, δημιουργούν ασφάλεια για τι επενδύσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, για την επίτευξη των στόχων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρθηκε από αρκετού σκιώδει ε, εισηγητέ. Χρειάζονται επενδύσει τη ΑΠΕ. Αυτό τι απαιτεί. Χρειάζεται συγκεκριμένε δεσμεύσει απο κάτι κράτη-μέλη να αυξηθούν οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσης και κρατών μελών. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πολιτικό πλαίσιο διαφανές στέρεο που δίνει βεβαιότητα για να προσελκύσουμε τι αναγκαίε επενδύσει. Αν δείτε ποια είναι η σημερινή κατάσταση που αναφέρει η έκθεση, ποια είναι η σημερινή κατάσταση, τι βλέπουμε. Ότι η παρούσα ενεργειακή πολιτική και η πολιτική για τις ΑΠΕ που στηρίζει την οδηγία 2009 είναι αποτελεσματικό εργαλείο. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουν στην πορεία που θα οδηγήσει σε στόχο για ΑΠΕ 20% ε, μέχρι το 2020. Σήμερα το μερίδιο των ΑΠΕ είναι στο 16%. Τα επίσημα στοιχεία είναι αυτά του Ευρωστάτ που αφορούν το 2014. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 27,5% ΑΠΕ στον τομέα ηλεκτρικής, 17,8% στη θέρμανση και ψήξη και 6% στις μεταφορές. Πράγματι, οι μεταφορές έχουν μείνει πίσω. Ελπίζουμε να καλυφθεί το κενό με την αναθεώρηση της οδηγίας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πρόοδος είναι καλή και όπως ανέφερε και ο συγγετής του ΕΛΚ, είμαστε σωστή πορεία. Μπορούμε να πούμε σωστή πορεία για την επίτευξη των στόχων του 2020. Τι βλέπουμε, ότι νέα κράτη-μέλη ήδη έχουν πετύχει τους στόχους. Τους εθνικούς τους στόχους του 2020, αλλά τρία κράτη-μέλη είναι σε καλή πορεία προς επίτευξη των στόχων του 2020, ακόμα και φέτος. Ο πρόεδρος. Α, και κάτι άλλο να πείτε. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη προχωρούν αρκετά καλά, βλέπουμε ομάδα κρατών μελών που χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια να πετύχουν τους στόχους του 2020 και τα επόμενα χρόνια. Είμαστε στενή επαφή με τα νοοκράτη κράτη-μέλη. Παρακολουθούμε το πώς προχωρούν. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε να επανεξετάσουν τους εθνικούς στόχους και στρατηγικές για τις ΑΠΕ και να εξετάσουν σοβαρά την χρήση μηχανισμών συνεργασίας που βρίσκονται στην οδηγία για τις ΑΠΕ. Επίσης σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι οι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι του 2020 δεσμεύουν τα κράτη-μέλη και θα επιβληθούν. Πέρα μετά το 2020 τι γίνεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει τις προτάσεις της, τις σχετικές. Θα τις υποβάλει πριν το τέλος του έτους, στα πλαίσια ευρυτέρου πακέτου, που αφορά επίσης την αναθεώρηση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αγορές θα γίνουν πιο ευέλικτες. Και έτσι θα υπάρχει καλύτερη ένταξη των ΑΠΕ. Θέλουμε να δούμε ποια μέτρα θα βοηθήσουν τα κρατημένη να πετύχουν από κοινού το 27% ΑΠΕ στο μείγμα. Θα λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, ψήξης και μεταφορών και θα δούμε με, καλύτερο, με καλύτερο τρόπο να δώσουμε τη δυνατότητα στους κατανοτές που θέλουν να παράξουν, να αποθηκεύσουν και να απολύσουν τη δική τους ενέργεια να το κάνουν και με τρόπους επίσης θα εξετάσουμε για να μειώσουμε το διοικητικό άχθος και τους φραγμούς και να δώσουμε και κίνητρα για να δημιουργηθεί εργατικό δυναμικό με τις κατάσταση εξώτηξης του τομέα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η κυρία Σιγήτρια έχει το λόγο. Τα τελικά σας σχόλια θέλουμε να ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όσους έλαβαν το λόγο και για το περιεχόμενο των ε, συμβουλών τους που ήταν τόσο χρήσιμες. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση καταρχήν. Γιατί να κατανομάζουμε τις χώρες. Η έκθεση αυτή προσπαθεί να, και εδώ απηχώ τα λόγια της Κομισιόν, να στοιχηματίσει υπέρ του υπέρ της βοήθειας κάποιων κρατών που ενδεχομένως θα έχουν πρόβλημα για τους στόχους το 2020. Το να κατανομήσουμε τους, χώρε τις χώρες αυτές βοηθά στο να βελτιώσουν αυτά τα οποία λαμβάνουν έτσι ώστε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας. Και χωρίς να θέλουμε να αμφισβητήσουμε το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, νομίζω ότι Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνται τα κράτη-μέλη και όντως στείλουν τους μηχανισμούς που θα τους επιτρέψουν να φτάσουν ε, στα αποθητά αποτελέσματα. Αναμφίβολα, αυτή η εξέταση αυτών των κρατών θα πρέπει να γίνεται δημοκρατικά και με σεβασμό για τους εθνικούς κανόνες. Αυτό που φαίνεται στην έκθεσή μας είναι πως οι στόχοι θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί, γιατί έχει αποδειχθεί ε, δε πως αυτό είναι το πιο λειτουργικό δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε εν ώψη του 2030 τα μέτρα να είναι λιγότερο φιλόδοξα από ό,τι οι στόχοι που είχαμε ορίσει για το 2020. Και αυτό συμπεριλαμβάνει οι στόχοι του 2020 να θεωρηθούν ως υποχρεωτικά υποχρεωτικά. Ε, εκπληρωτεί έτσι ώστε να είναι το κατάλληλο σημείο αφετηρία για την οδηγία που θα καλύψει την επόμενη περίοδο. Εν πάση περιπτώσει θεωρούμε πω είναι ουσιαστικό να έχουμε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα είναι σταθερό, θα είναι σίγουρο και το οποίο όντω θα στοιχηματίσει υπέρ των επενδύσεων Όπω επίση και των δημοσίων επενδύσεων ακριβώ ε, για να συνεχίσουμε να έχουμε επενδύσει σε αυτόν τον κλάδο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Είμαι πασιχαρούμενη που έλαβα τόσες πολλές τροπολογίες και όσες υπόλοιπε έρθουν και θα ξεκινήσω με όλες μου τις δυνάμεις να συνεργάζομαι και να ε, καταλήξω σε κάποιους συμβιβασμούς που θα επιτρέψουν σε αυτή την έκθεση να περάσει εύκολα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Συγήτρια. Θα τα ξαναπούμε στις 3. και έχουμε την ακρόαση εκεί με τον ανασχεδιασμό της ε, αγοράς, ε, της αγοράς ενέργειας. Θα τα πούμε λοιπόν σε 2,5 ώρες.